Monsieur le Président de la Αγαπητέ Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητέ κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε Γκουαλτιέρη της δικής μας Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς, ησυχία. Σιωπή παρακαλώ. Είναι μια συνεδρίαση εξαιρετικά σημαντική, δημόσια συνεδρίαση, Χαιρετώ το κοινό. Είναι μια συνεδρίαση που διαδίδεται διαδικτυακά και αυτό σημαίνει ότι όλος ο κόσμος έχει το βλέμμα του στρα... στραμμένο πάνω μας. Για λόγους που όλοι γνωρίζετε και καταλαβαίνετε, ξεκινούμε με λίγη καθυστέρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Γιούγκερ και τον επίτροπο Μοσκοβισή, διότι δέχθηκαν να παραμείνουν για 15 λεπτά παραπάνω Έχουμε όμως μισή ώρα καθυστέρηση και θα προσπαθήσουμε να διοργανώσουμε την συνεδρίαση ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε να πάρουν το λόγο όλοι οι ομιλητές που έχει προβλεφθεί να μιλήσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα ιδιαίτερο τον πρόεδρο Jean-Claude Juncker και πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι είναι πρεμιέρα η σημερινή εδώ και πάρα πολύ καιρό. δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ανατρέξει στις προηγούμενες εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρχει προηγούμενο σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εμφανίζεται ενώπιον δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνήθως ο πρόεδρος της Επιτροπής έρχεται στην Ολομέλεια και στην διάσκεψη των Προέδρων των πολιτικών ομάδων ή των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Σήμερα όμως έρχεται ενώπιον δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών και αυτό έχει να κάνει με τη σοβαρότητα του θέματος. Γνωρίζετε, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλησε να ε, κομίσει τη δική του πολιτική απάντηση στο σκάνδαλο LuxLeaks συστήνοντας την Ειδική Επιτροπή για προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και άλλα μέτρα παρεμφερή στη φύση ή στο αποτέλεσμα, την Επιτροπή TAX δηλαδή, η οποία να εργαστεί από κοινού με την Επιτροπή Οίκων Οικονομικών Υποθέσεων για να μελετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι συμβαίνει στα 28 κράτη-μέλη ε, σε ό,τι αφορά ε, τις διοικητικές ε, πρακτικές, ε, το φορολογικό δίκαιο και το πώς ωφελούνται ή δεν ωφελούνται οι επιχειρήσεις από το φορολογικό καθεστώς των χωρών. Και επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να υποβληθούν συγκεκριμένες προτάσεις. Αντιστοίχως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιδράσει πολύ γρήγορα με τη σειρά τη και από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είμαστε σε φάση σύνταξη της έκθεσής μας και θα έχουμε τα τελικά συμπεράσματα, επιθυμούμε να έχουμε και την παρουσίαση της άποψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την παρουσίαση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό. Εξού και έχουμε μαζί μας τον Επίτροπο Μοσκοβισή, αλλά και στη συνέχεια θα ε, κάνουμε ακρόαση της Επιτρόπου Φεστάγκερ. Και θα έχουμε έγγραφα από τα λοιπά θεσμικά όργανα κύριο μέλημά μας είναι, και τελειώνω με αυτό το μήνυμα, είναι η διατήρηση της άσκησης πολιτικής πίεσης. Κύριο μέλημά μας είναι να κινηθούμε το, όσο το δυνατόν ταχύτερα έτσι ώστε ε, να υιοθετηθεί από τα 28 κράτη-μέλη το σχέδιο απαραίτητων μεταρρυθμίσεων επί τη βάση των προτάσεων που θα έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και τις οποίες θα ενσωματώσουμε σε μεγάλο βαθμό στην έκθεσή μας. να πω παρεθετικά ότι χρειάζεται ομοφωνία από πλευράς κρατών μελών για το θέμα αυτό. Να δώσω το λόγο στον πρόεδρο Γκουαλτιέρη, ο οποίος θα προεδρεύσει κατά το ίμιση της συνεδρίασης και δεδομένου του ότι ο χρόνος πιέζει, σας προτείνουμε να έχουμε δύο γύρους παρεμβάσεων. Ένα πρώτο γύρο που θα επιτρέψει στον εκπρόσωπο της κάθε πολιτικής ομάδας να πάρει το λόγο, ε, όχι περισσότερο από δύο λεπτά ο καθένας και στη συνέχεια να υπάρξει η απάντηση από τους παριστάμενους. Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Αλέν. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον Πρόεδρο Γιούνκερ και τον Επίτροπο ε, Μοσκοβισή που έχουν έρθει που δέχτηκαν αυτή τη τόσο σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ ήδη συνεργάζεται εξαιρετικά με την Επιτροπή ΤΑΞ. Κάνουμε εξαιρετικά σημαντική και καλή δουλειά. Από τη δική μας πλευρά εργαζόμαστε από, επί της νομοθετικής πλευράς των υποθέσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει ε, στην εξετασή τους μέσω της αυτόματης ανταλλαγής απόψεων και ανέκαθεν, εκτιμούσα πολύ ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι η Επιτροπή του είναι πολιτική επιτροπή. Ε, είναι νέο, είναι μεγάλη και σημαντική συνταγματική εξέλιξη και πιστεύω πως ε, έτσι ε, θετικά επηρεάζει αυτή η κατάσταση, τη σχέση που νομίζω πως θα έπρεπε να έχουμε νομοθετικά στο έργο του Κοινοβουλίου και στη συνεργασία με την Κομισιόν. Εγώ καλωσορίζω το πρόγραμμα δράσης, όπως δείτε έχουμε ήδη ένα σχέδιο και μια ακόμα πιο φιλόδοξη πρόταση και βεβαίως αναμένουμε η Κομισιόν να τα λάβει όλα αυτά σοβαρά υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα ξεκινάμε την συνεδρίαση με τον πρόεδρο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ. Μάλιστα κύριε πρόεδρε. Κυρία εισηγήτρια, κύριε εισηγητά, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, αγαπητέ επίτροπε. Ο πρόεδρος Λαμασούρη είπε ότι δεν ήθιστε ο πρόεδρος της Επιτροπής να παρουσιάζεται, όχι βέβαια σε αυτό του είδους τη αίθουσης, αλλά πιστεύω πως είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί είχα πει ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής θα ήταν ανάμεσα στις προτεραιότητες της Επιτροπής αυτής και άρα και του Προέδρου της. Είναι απόλυτα φυσιολογικό λοιπόν ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Επίτροπος επί της αρμόδιος για τα φορολογικά θέματα να παρουσιάζονται ενώπιόν σας. Όντως ε, η Κομισιόν της οποίας προεδρεύω έχει τοποθετήσει την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροαπάτης ε, μέσα στις 10 πρώτες της προτεραιότητες ε, γιατί θέλουμε πραγματικά να την καταργήσουμε τη φοροαπάτη στη αποφυγή και φοροδιαφυγή. Πιστεύουμε ότι η Ένωση και η Ενωμένη Αγορά είναι ατελείς εφόσον υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί η εσωτερική αγορά εκεί όπου δει και συγκεκριμένα στα θέματα φορολογίας και φορολόγησης και αυτό σημαίνει φορολόγηση εταιριών και θέλουμε με σταθερό βήμα να προχωρήσουμε σε περισσότερο ε, συντονισμό και ε, συγχρονισμό. Είναι ένα είδος δοκιμασίας για να δούμε κατά πόσο θέλουμε να συνδυάσουμε, συμβιώσουμε με, συγχωρείτε, σε, με συγκεκριμένους και συμπεφωνημένους όρους. Ως ε, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτοί που ήδη σκογελάνε εκεί πέρα, αυτοί οι δυο πρασινούλιδες που είναι μπροστά μου, ξέρουν πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω, γιατί τα συζητήσαμε μαζί ε, όταν είχα άλλη ιδιότητα. Δεν ανακαλύπτω λοιπόν το θέμα το φορολογικό, διότι όταν ασκούσα το λειτουργήμά μου στην χώρα μου, ε, είχα αναλάβει αυτά τα θέματα. Θα σας το θυμίζω, αλλά θα το γνωρίζετε ήδη, ότι όταν προείδρευα το 91 του Συμβουλίου ε, ΕΚΟΦΗΝ, πριν από 24 χρόνια, ήμουν νέος Υπουργός ε, Οικονομίας τότε και είχα καταφέρει να πείσω τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν το ΦΠΑ και τους ειδικού φόρους κατανάλωσης στην Ευρώπη με πολύ ισχυρή βούληση που εμπνεύστηκε από μάλλον έναντι πολύ ισχυρή βούληση που νεότερα από αντίθετε απόψει. Οι Βρετανοί έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να ασχολείται με τα θέματα φορολογία γιατί αυτή υπόκειται στον κανόνα της ομοφωνίας. Δεν έλεγαν οι Βρετανοί, ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Επίσης το 1997 ήμουν υπουργό Οικονομικών όταν φτάσαμε τον κώδικα διοντολογίας κατά της, του αθέμητου ανταγωνισμού ανάμεσα στις εταιρείες και επίσης φτιάξαμε και την εναρμόνιση της φορολόγησης των αποταμιεύσεων στη συνέχεια. Θα σας θυμίσω, αλλά και αυτό επίσης το ξέρετε, ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΕΚΟΦΗΝ, ε, πρότεινα, τη δημιουργία μιας φορολογικής επιτροπής, γιατί θεωρούσα ότι τα θέματα τα φορολογικά έχουν την ίδια σημασία όπως και τα ε, νομισματικά και τα οικονομικά. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου, προεδρεύων του Συμβουλίου το 2005 δεν τα κατάφερα. Δεν θυμάμαι πια ποιες κυβερνήσεις ήταν υπέρ, ποιες ήταν κατά. Δεν θυμάμαι Θυμάμαι όμως ε, την στήριξη του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και επανέφερα αυτήν τη συζήτηση στις προπαρασκευαστικές συζητήσεις που μας οδήγησαν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, επανέφερα το θέμα δεν θυμάμαι ποιοι ήταν υπέρ και ποιοι ήταν κατά τότε, αλλά δεν τα καταφέραμε ούτε τότε. Πάντως το ξαναλέω τώρα πως εάν θέλουμε το ευρωπαϊκό, ε, η ευρωπαϊκή φορολόγηση να έχει την ίδια σημασία όπως και τα υπόλοιπα θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα της δημιουργίας μιας ε, φορολογικής επιτροπής ε, που θα παρακολουθεί τις εργασίες της ομάδας για τον κώδικα δεοντολογίας και που θα εμπνέει στη συνέχεια τις εργασίες των Υπουργών Οικονομικών. Είμαι βέβαιος ότι θα συγκρατήσετε αυτή την ιδέα που είναι απλώς κοινή λογική. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και στη στιγμή που έπρεπε να παρουσιάσω τους δικούς μου πολιτικούς προσανατολισμούς καταρχήν και μετά αυτούς της Κομισιόν, ανέκαθεν έθετα ε, την έμφαση στην ε, καταπολέμηση της ε, φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και είπα και πέρυσι ότι θα αποδώσουμε την απαραίτητη ε, προτεραιότητα στις στατικικές βέλτις της ε, φορολόγησης των πολυεθνικών εταιριών. Η Κομισιόν έχει διάφορες, έχει μάλλον ξεκινήσει διάφορες διαδικασίες κατά ορισμένων κατορμελών όπως η χώρα μου και ε, πόσο γνωρίζω, εξ όσο γνωρίζω, ε, συνεχίζονται οι σχετικές διαδικασίες. Υπό το, την Επίτροπο Βεστάγκερα που είναι ειδικό και που έχει αναλάβει το θέμα και έχει μεγάλη αυτονομία. Δεν χρειάζεται ούτε τις δικές μου υποδείξεις, ούτε παροτρύνσεις, ούτε συμβουλές, διότι ε, γνωρίζει πάρα πολύ καλά το θέμα. Δεν ανακατεύομαι καθόλου σε αυτές τις διαδικασίες και δεν χρειάζεται και να ανακατευτώ διότι η Επίτροπος αυτό που είναι αρμόδια για την, ε, τον ανταγωνισμό έχει μεγάλη αυτονομία. Εκ... Ούτως ή άλλως έπρεπε να απέχω διότι πρόκειται για τη χώρα μου. Άρα για, για προφανή διοντολογικούς λόγους έπρεπε να απέχω από όλη αυτή τη διαδικασία. Κατά τα λοιπά όμως έχω υποχρέωση ε, δράσης. Ε, και εγώ και ο Επίτροπος Μοσκοβισή. Πρέπει να ενεργήσουμε. Από τη μια πλευρά απέχω τη διαδικασία, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ενεργήσω. Δεν θα πρέπει να αμφιβάλλεται για τη βούλησή μας να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε στον συντονισμό και στην εναρμόνιση. Και στην εναρμόνιση. Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα ειδικών προνομιακών φορολογικών καθεστώτων, tax rulings. Έχουμε Υποβάλλει αυτή την πρόταση, την επέβαλε ο Πίτροπο Μοσχοβησή και πιστεύω πω η Πορτογαλική, η, συγγνώμη, η Προεδρία του Λουξεμβούργου θα προχωρήσει στην υιοθέτηση αυτή τη απόφαση μέσα στον Οκτώβριο. Δεν είναι κακό αυτό γιατί δίνει στον επιχειρηματικό κόσμο μια δυνατότητα προβλεψιμότητας για την οποία οι οικονομικοί φορείς τη χρειάζονται. Tax rulings λοιπόν απόφαση προκαταβολική είδαμε τα λάθη του παρελθόντος και τις αρνητικές επιπτώσεις όταν δεν είναι αρκετά καλά πλαισιωμένος ένας χώρος. Γι' αυτό και θέλαμε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Είχα αναπτύξει αυτή τη θέση μου και ενώπιόν σα. Είχα αναπτύξει τη συνεδρίαση ε, το στο Brisbane οι υπόλοιποι δεν το δέχτηκαν με τεράστιο ενθουσιασμό, αλλά και εκεί χρειάζεται να υπάρξουν καθολικές συμφωνίες. Αν δεν καταφέρουμε να πείσουμε τους εταίρους του G20, εμείς θα το κάνουμε στο επίπεδό μας και για τα δικά μας, ε, τις δικές μας εταιρείες. Είχαμε πει ότι θα ε, προχωρούσαμε έτσι ώστε σε θέματα φορολόγησης επιχειρήσεων να έχουμε κοινούς κανόνες για το, τη, τη βάση φορολόγησης και, και από αυτό εργαζόμαστε. Ταυτόχρονα η ανάγκη για ανάπτυξη, η ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις, δεδομένου ότι λείπουν οι επενδύσεις αυτή τη στιγμή, η ανάγκη να αφαιρεθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη της απασχόλησης Πιστεύουμε πως η φορολογία των επιχειρήσεων δεν πρέπει να αποτελεί φρένο σε αυτή τη γενική προσπάθεια ανάπτυξης. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί, όπως έλεγα, να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά. Το σύστημά μας αυτή τη στιγμή είναι δυσνόητο και άδικο. Υπάρχουν αυτοί που χάνουν λόγω αυτής της αδικίας και της ε, ε, ασυνεννοησίας, αλλά υπάρχουν και αυτοί που, χα, που κερδίζουν, γιατί μπορούν να κρυφτούν πίσω από την ποικιλομορφία των εθνικών νόμων που καθιστούν το τοπίο ε, σκοτεινό και αδιαφανές. Πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των μεγάλων επιχειρήσεων που θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι χαίρουν ε, μεγάλης φορολογικής ευελιξίας ε, και ικανότητας. Εκμεταλλεύονται κάθε φορά τις διαφορετικές εθνικές φορολογικές ε, πρακτικές. Και πρέπει λοιπόν να βάλουμε τάξη γιατί όλα αυτά οδηγούν σε άδικες συνέπειες σε αυτό το πεπαλαιωμένο σύστημα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα για τα οποία μιλάω, γιατί ο κόσμος έχει γίνει παγκόσμιοποιημένος, η οικονομία, η ψηφιακή έχει γίνει ε, κινητή και θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε τα κράτη-μέλη να φτιάξουν και πολύ πιο στενή συνεργασία σε αυτά τα θέματα από ό,τι αυτοί που έχουν ε, μέχρι τώρα. Καθώς επίσης, επειδή παρατηρούμε, και είναι καλό αυτό το σημείο, ότι υπάρχει μια γενική κινητοποίηση για την καταπολέμηση των φορολογικών απατών. Άρα λοιπόν κοινή φορολογική βάση ε, είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μια κοινοτική μέθοδο για να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα των PEPS. Είμαστε όλοι κομμάτι της ε, κοινής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να έρθουμε στο ίδιο επίπεδο να ευθυγραμμίσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εναρμόνιση φορολογική δεν σημαίνει το πέρας ενός υγιούς φορολογικού ανταγωνισμού, δηλαδή να θέλουμε να φτιάξουμε καλούς, απλούς και αποτελεσματικούς κοινούς κανόνες ε, ε, ώστε να μην υπάρχει αθέμητος φορολογικός ανταγωνισμός. Γι' αυτό και με τον Ζαμπιέρ προετοιμάσαμε προτάσεις που βασίζονται σε κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Οι, τα κέρδη θα πρέπει να φορολογούνται στη χώρα όπου δημιουργούνται. Και η δεύτερη αρχή, η κατευθυντήρια αρχή, είναι να μην ξεχνάμε ότι τα η πολιτική, η φορολογική θα πρέπει να στηρίζει την πολιτική απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και ο μόνος τρόπος για την μείωση του κόστους συμμόρφωσης είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα εγγυάται την νομική ασφάλεια και βεβαιότητα, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει και να απογειωθεί. Είναι πολύ σημαντικό να φτάσουμε γρήγορα σε ανταλλαγή απόψεων σε μάλλον αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στα θέματα ε, των tax rulings, γιατί έχουν αυτά διαμεθοριακή επίπτωση είναι ένας από τους βασικούς άξονες ε, που εμπεριέχεται στα όσα είπε ο Επίτροπος ε, Μοσκοβιστή τον περασμένο Ιούνιο όταν παρουσίασε το πλάνο δράσης, όταν είπαμε Εξάλλου ο Πιέρ θα σας εξηγήσει με λεπτομέρειες αυτές τις φιλοδοξίες. Εγώ δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για αυτά τα θέματα, θα πω μόνο ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες για θέματα της κοινή πλατφόρμας φορολόγησης για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ο κ. Μοσκοβισή παρουσίασε ένα σχέδιο σε, διάφορες, ε, σε διάφορα στάδια. Θα πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και εδώ μεταξύ να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε για κάποιες αρχές ε, κοινέ ώστε αυτή η αταξία να διορθωθεί. Ο πρόεδρος αλλά μου λέει πως ήδη εξήντλησα το χρόνο μου. Το δέχομαι. Γιατί θα ήθελα να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Αν αμφίβολα έχετε ερωτήσεις για τα διάφορα θέματα του Λίλξ ε, και βεβαίως δεν θέλω να σας τηρήσω τη χαρά να τα υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Thank you. ευχαριστώ. Πρόεδρε, Πρόεδρε. Jean-Claude Juncker. Και τώρα το λόγο δίνω στον Πιέρ Μοσκοβιστή. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου, όπως και ο πρόεδρος Γιούγκερ το έκανε, γιατί το σχέδιο έκθεσης είναι εξαιρετικά καλό και πολλά στοιχεία του είναι ευπρόσδεκτα για εμάς. Μας εμπνέουν για τη συνέχιση των εργασιών μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας προτεραιότητα, μία από τις προτεραιότητες είναι η φορολογία. Πρόκειται για μία επανάσταση, για μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ε, απλούστευση. Δεν θέλω να μακρηγορήσω θα ήθελα ε, σε λίγα λεπτά να μιλήσω για το AXIS, το CCCTB, την φορολογική διαφάνεια και την πραγματική φορολόγηση. Πρώτον, ως προς το AXIS, την ενοποιημένη κοινή φορολογική βάση για τον ε, φόρο επί των εταιριών. Χαίρομαι διότι το project αυτό, το έργο αυτό έχει ε, νέα ορμή βρίσκεται στο τραπέζι του Συμβουλίου Υπουργών χωρίς συμφωνία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εάν όμως προχωρήσουμε βήμα-βήμα, στάδιο-στάδιο, τότε θα προχωρήσουμε καλύτερα και περισσότερο. Ο ρεαλισμός επιτάσσει να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, να μην χάσουμε την ενοποίηση από τον όραμά μας και από τον ορίζοντα, αλλά ας μην πάμε μέχρι εκεί σε πρώτη φάση, ας πάμε στην κοινή φορολογική βάση. Και υπάρχει και το έργο BEPS, η καταπολέμηση δηλαδή της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών, των ενδομιλικών συναλλαγών δηλαδή. Θα έχουμε τον ορισμό της έρευνας και της ανάπτυξης μεταξύ άλλων και θα ε, ασχοληθούμε με τα πιο σημαντικά ε, θέματα όπως είναι και η ε, χρέωση, η δημιουργία χρεών από πλευράς επιχειρήσεων. Το Axis είναι το καλύτερο εργαλείο για να έχουμε αποτελέσματα και σε θέματα διαφάνειας και σε θέματα αποτελεσματικότητας και γι' πρέπει να συντάξουμε μια αναθεωρημένη πρόταση ποιοτική που θα δώσει νέα ορμή στι διαπραγματεύσεις των κρατών μελών οι οποίε είναι αρκετά ασθενεί αυτή τη στιγμή. Ω προ τη φορολογική διαφάνεια και το reporting την υποβολή αναφορά αναπεπραγμένα χωρών, αναχώρα. Η δική σας Επιτροπή ενδιαφέρεται ιδιαίτερως γι' αυτό. Για τη διαφάνεια λοιπόν χαίρομαι διότι το σχέδιο έκθεσή σας στηρίζει την πρόταση οδηγίας για τα tax rulings, τα ειδικά προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και θα είμαι και πιο συγκεκριμένος. Μετά το τελευταίο τελευταίο συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ το άτυπο στο Λουξεμβούργο επιθυμώ ε, το κείμενο να εγκριθεί στο επόμενο ΕΚΟΦΗΝ στις 6 Οκτωβρίου για να αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2016. Δεν θα είναι αποδεκτό η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πρόδρομος και πρωτοπόρος όλα αυτά να φτάσει μετά ε, τον ΟΣΑ, ε, δεύτερη και καταϊδρωμένη. Μετά τον Περί Pain έχει γίνει πολλή δουλειά. Στην Άγκυρα έχει ήδη γίνει λόγος ε, για το θέμα αυτό και για μια κοινή βάση. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου και υπάρχουν αλλά είμαι σίγουρο ότι θα καμφθούν. Μία δεύτερη κόκκινη γραμμή δική μα είναι η εξή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να είναι ε, συμβαλόμενο μέρο και αναπόσπαστο μέρο του μηχανισμού θα διασφαλίσει ότι οι πληροφορίε πράγματι ανταλλάσσονται μεταξύ των χωρών μελών. Γνωρίζετε την προσωπική μου προτίμηση, δεν την κρύβω, το λέω και ξεκάθαρα. Μιλούμε για να γίνει ε, η δημοσίευση και η δημοσιότητα των στοιχείων αναχώρα πραγματικότητα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτό το οποίο μας επιτάσσει η οικονομική αποτελεσματικότητα, που μας επιτάσσει η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο συνάδελφος Χιλ, ο Επίτροπος Χιλ έχει προχωρήσει στο δικό του χαρτοφυλάκιο και στη συνέχεια θα πρέπει να συμφιλιώσουμε αυτές τις δύο απαιτήσει για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και στο χαρτοφυλάκιο Χιλ και στο χαρτοφυλάκιο το δικό μου Μοσκοβισή. Και έτσι ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συγκυρία στην Ευρώπη. Θα είμαστε αποτελεσματικοί. Επενδύσεις χωρίς διαφάνεια δεν θα είναι αποτελεσματικές και δεν θα κερδίσουν την εμπιστοσύνη του ε, πολίτη. Χαίρομαι διότι η Επιτροπή σας δρά για να έχουμε αποτελεσματική φορολόγηση των κερδών που υλοποιούνται και δημιουργούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί τίνος πρόκειται. Να αρνηθούμε δηλαδή μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία επιχειρήσεις δημιουργούν κέρδη, δημιουργούν πλούτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν λαβή για, ελάχιστο, ε, για ελάχιστη φορολόγηση ή και καθόλου φορολόγηση εκεί όπου δρούν. Υπάρχει το σύστημα της μη διπλής φορολόγησης. Αυτό το παραδεχόμαστε και καλώς, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε και σε ένα σύστημα που να έχουμε αποφυγή της διπλής μη φορολόγησης, δηλαδή να μην φορολογούνται ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Και υπάρχουν διάφορες παρανοήσεις Μιλούμε για αποτελεσματική λειτουργική φορολόγηση. Επί της ουσίας, στο ΕΚΟΦΗΝ είπα ότι η ομάδα πρέπει να τροποποιήσει τα κριτήρια για να δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην πραγματική φορολόγηση και ως προς τις ε, φορολογικές δικαιοδοσίες των τρίτων χωρών. Χαίρομαι γιατί η Επιτροπή σας στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήταν πολύ χρήσιμες οι εργασίες σας. Σας κριτήκαρα να απαντώ τόσο το καλύτερο γιατί σκοπός του καταλόγου είναι ακριβώς να βγει στην επιφάνεια και να τροποποιήσει τροποποιηθούν Θα προχωρήσουμε πέρα από τον ενοποιημένο κατάλογο που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο και αυτό που προτείνω είναι να συμπεριλάβουμε την εκπόνηση κοινών κριτηρίων και κυρώσεων. Δηλαδή, οι δικαιοδοσίε φορολογικέ και διοικήσει φορολογικέ τρίτων χωρών που δεν συνεργάζονται να υπάρχει διαφάνεια αλλά και κυρώσει. Βεβαίω πρόοδο δεν μπορεί να σημειωθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Όμω κάνουμε το παν για να σημειώσουμε πρόοδο ε, πάνω στην εξέταση όλων αυτών των θεμάτων που είναι περίπλοκα, που συνεχίζουν να εντάσσονται στον κανόνα τη ομοφωνία, ο οποίο είναι εξορισμού περιοριστικό. Και έχω την αίσθηση ότι ο Επίτροπος αρμόδιο για τα θέματα αυτά έχει την πλήρη στήριξη του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του συνόλου του σώματο ε, της έχουμε ομαδικό πνεύμα, σέβεται ο καθένας τη δουλειά του άλλου και εγώ τη δουλειά της Επιτρόπου Φεστάγκερ και αντιστρόφως, προχωρούμε, ωστόσο πρέπει να υπογραμμίσω ότι χωρίς πολιτική βούληση δεν θα υπάρξει αλλαγή και γι' αυτό η δική σας έκθεση και γι' αυτό η δική σας στήριξη και γι' αυτό η δική σας παρέμβαση είναι εξαιρετικά σημαντικές και θα το πω ξεκάθαρα και με αυτά κλείνω, χαιρετίζω με θέρμη την πίεση που ασκεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ειδική επιτροπή σας τάξε για προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και άλλα μέτρα παρεμφερεί, την πίεση που ασκείται στα κράτη-μέλη γιατί πραγματικά τη χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτροπή μας Και ιδιαίτερος για τις τελευταίες κουβέντες σας. Να ξεκινήσουμε με το γύρο των απαντήσεων. Θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ αυστηρό σε ό,τι αφορά το χρονικό όριο. Δύο λεπτά για κάθε ερώτηση. Κύριε Μπάλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, κύριε Επιτροπέ, σα ευχαριστούμε ιδιαίτερα που σήμερα ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μα. Και στι ε, δύο επιτροπέ ε, αυτέ, μάλλον. Ε, το εκτιμούμε ιδιαίτερα αυτό. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση από την πρακτική μου εμπειρία και από τη ζωή μου ως Ευρωβουλευτής έχω να θίξω κάτι. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής να σας πάρω μαζί μου σε μια επίσκεψη σε μια μικρομεσαία επιχείρηση στη Γερμανία, στο Λουξεμβούργο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την επίσκεψη λοιπόν ε, συζητάμε και ο επιχειρηματίας στρέφεται προς εσάς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας απευθύνει το εξής ερώτημα. Κύριε Γιούνκερ, γιατί οι μικρές επιχειρήσεις, οι μεσαίες, οι μεσαίοι επιχειρηματίες στις χώρες τους εξακολουθούν να πρέπει να τηρούν τις φορολογικές τους ε, υποχρεώσεις, ενώ οι πιο πολλοί πολυεθνικοί όμιλοι έχουν τη δυνατότητα να μηδενίσουν το φορολογικό τους φορτίο. Γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν τόσο λίγα ελάχιστα πρότυπα, όπως για παράδειγμα αυτά που αναφέρατε για την βάση υπολογισμού της φορολογίας των ε, ε, συνεταιρισμών, των ενώσεων και γιατί δεν υπάρχει κάτι γνωστό σε ό,τι αφορά τους μεγάλους παίκτες, τις μεγάλες επιχειρήσεις ανά χώρα, γιατί δεν αναφέρονται αυτά στην συγκεκριμένη έκθεση. Και έτσι λοιπόν ε, θα ήθελα να μου πείτε τι θα απαντούσατε συγκεκριμένα σε αυτόν τον άνθρωπο, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η κυρία Φεραίρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πορτογαλικά. Ως εισηγήτρια, μάλλον μια από τις εισηγήτριες, θα πρέπει να σας πω ότι διαπιστώνουμε ότι όχι μόνο επιβεβαιώνονται οι κατηγορίες και οι πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν στο LuxLeaks, αλλά πρόκειται για γενικευμένη πρακτική στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν δεν είναι πλέον δυνατόν να έχουμε μια ε, ένα ενιαίο νόμισμα, μια δημοσιονομική πολιτική κτλ. και ορισμένες χώρες να έχουν ε, ε κατά σύστημα να ζητούν μάλλον ε, φοροαπαλλαγές στις άλλες χώρες. Τώρα δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε καταγγελίες και να ρίχνουμε κατηγορίες ο ένας τον άλλον, αλλά θέλουμε να οργανώσουμε μια συγκεκριμένη προτεραιότητα ώστε να καλύψουμε αυτά τα κενά. Ε, για εμείς θέλουμε να πιέσουμε, να πιέσουμε πολιτικά αυτούς που μπλοκάρουν αυτό το θεματολόγιο. Εμείς χρειαζόμαστε πληροφορίες όμως γι' αυτό και στη διάρκεια των εργασιών μας αντιμετωπίσαμε μια μυστικοπάθεια που είναι βασικό χαρακτηριστικό για να μην προχωράνε τα πράγματα. Ο πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής ανέφερε τη δεκαετία του 90. Τη δεκαετία του 90 υπήρξαν προοδοί και ο ίδιος ο κώδικας διοντολογίας είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού. Αλλά είναι αλήθεια ότι από τότε δημιουργήθηκε αυτή η άγρια ζούγκλα στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Πώς εμείς λοιπόν να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση στην Κομισιόν για να συνεχίσει με αυτή την ατζέντα, αλλά και στα κρατημέλη, ώστε τα οποία μάλλον βολεύονται πίσω από το επιχείρημα της ομοφωνίας και έχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα ε, να υπερασπίσουν, αν δεν έχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρόσβαση σε πληροφορίες. Λούκε. Κύριε Γιούνκερ, αυτή η Επιτροπή δημιουργήθηκε γιατί με σκανδαλώδη τρόπο αποδείχθηκε ότι υπάρχουν ε, αποδεκτικά στοιχεία σε ως σχέση με φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή των μεγάλων ε, ομίλων. Ενδεχομένω νόμιμα. Η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να δράσει σε προλογικά ζητήματα, άρα ε, πήραμε τον πίσω δρόμο, αν θέλετε, με το Επικουρικό Δίκαιο, το οποίο και χρησιμοποιήσαμε για την βάση εργασίας της Επιτροπής. Δεν έχουμε συζητήσει όμως την Επιτροπή κατά πόσον ε, πρόκειται για ε, παράνομες ε, κρατικές επιδοτήσεις. Δεν το συζητήσαμε. Σας ζητώ όμως ε, από εσάς, γιατί σε εσάς εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και το πεδίο της εντολής σας. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον για να δεσμεύσει τις επιχειρήσεις αυτές που επιλέγουν αυτή την απαλλαγή από το φορολογικό καθεστώς. Είναι η αντίφαση τεράστια. Αφενός έχουμε ε, μια σαφέστατα εθνική αρμοδιότητα της ε, φορολογικής ρύθμισης και της ευρωπαϊκής ρύθμισης από την άλλη της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας για την ρύθμιση της ιστορικής αγοράς όπου συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των επιδοτήσεων. Πώς μπορεί να επιληθεί αυτή η αντίφαση δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιλέξει την προσέγγιση της φορολογικής εναρμόνισης. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος αλλά, εν πάση περιπτώσει, να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Θα ήθελα όμω να μα πείτε τι θα κάνετε κατά των παράνομων επιδοτήσεων, δηλαδή φορολογικέ, ε, μάλλον χρηματικέ ελαφρύνσει που δεν είναι άδικο πλέον έκτημα στον ανταγωνισμό σε μια επιχείρηση. Πιστεύετε, πιστεύετε όπως και εγώ, ότι σε κάθε περίπτωση η μετεγκατάσταση μιας εταιρεία σε μια διαφορετική δικαιοδοσία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ε, εξετάζεται και κλείνει δυστυχώς το μικρόφωνο ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Στόιρερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι πάρα πολύ σημαντικό που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Η φορολογική πολιτική στην Επιτροπή μας είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε για να δούμε τι γίνεται με τις επιχειρήσεις και τους μεγάλους ομίλους που επωφελούνται από τα παραθυράκια. Αυτό είναι συνήθις πρακτική. Αυτές οι πρακτικές υπονομεύουν τη φορολογική βάση άλλων κρατών μελών και επίσης ε, οι πολίτες, οι κανονικοί πολίτες και οι μικρές επιχειρήσεις δεν ωφελούνται από αυτό το όφελος. Εσείς μιλήσατε για την θητεία σας ε, ω Υπουργός στο Λουξεμβούργο. Υπάρχει μήπως μια ανίερη συμμαχία μεταξύ των μεγάλων ε, ομίλων και των μεγάλων επιχειρήσεων συμβουλευτικής ε, ω και ε, κυβέρνηση. Μπορείτε να θεωρήσετε ότι έχετε κάποια αρμοδιότητα ή είσαστε αβοήθητοι. Και κοιτώντας τι έγινε στο LuxLeaks. Ποιος εφήβρε το σύστημα αυτό, το ανεχτήκατε ήταν οι επιχειρήσεις αυτές οι οποίες το κυνήγησαν, ήταν οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις ή και οι τρεις παράγοντες. Ύστερα, εδώ και 20 χρόνια στις συνόδους συζητιόνται τα προβλήματα με τις πρακτικές ορολογικής αποφυγής ε, από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Το συζητούσαμε όμως μόνο. Γιατί δεν επιλύθηκε το πρόβλημα. Ποιος μπλόκαρε το ζήτημα αυτό. Γιατί σε σημαντικά ζητήματα ξέρουμε αν είμαστε υπέρ ή κατά. Υπάρχουν πρακτικά. Στα πρακτικά πρέπει να φαίνεται ποιο έκανε τι. Πότε θα μα τα δώσετε λοιπόν αυτά τα πρακτικά, αν είσαστε υπέρμαχο ε, των, ε, αν είσαστε όντω υπέρμαχο τη εξέβρεση λύσεων, θα πρέπει ω δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο να απαιτήσουμε αυτά τα έγγραφα και δεν ε, δεχόμαστε το ότι δεν μα τα χορηγούν. Και πραγματικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τώρα το ζήτημα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ο Φάμπιο Ντεμάζη. <coughs> Κύριε Γιούγκαρε, ο δημοσιογράφο από το Λουξεμβούργο Λεωνίκη του Ζουλμπουζό θέλει ότι, ότι ο κύριο Κρέκη, στην έκθεση Κρέκη, ε, ότι έχουν αφαιρεθεί κάποιες σελίδες οι οποίες θεωρούνταν πάρα πολύ επικίνδυνες για το Λουξεμβούργο και σε ό,τι αφορά το κοινωτικό δίκαιο και σε ό,τι αφορά τα tax rulings. Και ότι αυτό δεν το έχει αρνηθεί η κυβέρνηση ε, του Λουξεμβούργου. Κυρία Μπουζόλ, ε, διατείνεται ότι τις έχετε στις αυτές τις σελίδες η δημοσιογράφος κυρία Μπουζόλ. Λέει η αλήθεια. Λοιπόν, η κυρία Μπουζόλ και θα μας υποστηρίξετε στην περίπτωση αυτή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να πάρουμε και τις υπόλοιπες σελίδε και να έχουμε έτσι όλη την έκταση Κρέκελ. Δεύτερον, ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Αληθεύει ότι τα Χριστούγεννα όταν ε, είχατε ευθύνε και αξίωμα στο Λουξεμβούργο είχατε συναντηθεί με τον πρώην διευθυντή της ε, Commerzbank και της ε, ότι συναντηθήκατε και συζητηθήκατε και συζητήσατε το φορολογικό καθεστώς και τη φορολογική επιβάρυνση της ε, Commerzbank. Αν αυτό αληθεύει, πώς το αξιολογείτε α, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά το καθεστώς για τις ε, Ο Λαμπαγά, ένας ε, δημοσιογράφος στο Λουξεμβούργο, ε, το Παγκέλ διώκεται και ποιο είναι το καθεστώ, πείτε μα, σε ό,τι αφορά του whistleblowers, του πληροφοριοδότε, δεδομένου ότι η Επιτροπή δημοσίευσε προτάσει που μειώνουν την προστασία των πληροφοριοδοτών. Ευχαριστώ. Ο Σβέν Γκίγκολτ. Uh, Πρόεδρε, από τότε που αναλάβατε το 1989 το μερίδιο των κερδών των ΗΠΑ μέχρι το τέλος της δικής σας εντολής στο Λουξεμβούργο από το 0 ε, στο 89, το 1989 έχει ανέλθει στο 10% σήμερα. 10% ξένες, ε, ξένα κέρδη ε, είναι αυτά. Είστε έτοιμος να πείτε ε, συστηματικά ποιο ρόλο παίξατε εσείς στη δημιουργία του φορολογικού παραδείσου του Λουξεμβούργου. Δεύτερον, εσείς ε, καθιστάτε την διαφάνεια ως προτεραιότητα της ε, Προεδρίας σας και το κάνετε. Ωστόσο η Κομισιόν σας δεν μας έδωσε τα έγγραφα για τον κώδικα, για τον κώδικα του διοντολογίας για να, που είναι κρίσιμα για να καθορίσουμε ποιος έλαβε ποια θέση ώστε να πάψουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να ε, επιτρέπουν τον αθέμητο ανταγωνισμό στη φορολογία. Μιλάμε για τουλάχιστον 500 σελίδες πρακτικών από τις βασικές συνεδριάσεις από το 1988 και την προσπάθεια που έχει κάνει η υπηρεσία σας για τις συνθήκες του TTIP ε, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει, δεν μπορούμε να κρατάμε σημειώσεις, δεν μπορούν να κρατάνε σημειώσει, ενώ πρόκειται για πολύ τεχνικά ζητήματα. Θα μας δώσετε τα έγγραφα, διότι αυτοί οι κανόνες για πρόσβαση στα έγγραφα πραγματικά ε, δυστιμούν τη δημοκρατία. Και άλλο ένα σημαντικό ερώτημα για μένα είναι, αν τα έγγραφα αυτά δεν δημοσιοποιηθούν, στην Επιτροπή μας ή τουλάχιστον υπό κάποιες ε, σοβαρές προϋποθέσεις να είναι διαθέσιμα, δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε την εντολή μας και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να μπορούμε να παρατείνουμε αυτή την εντολή γιατί διαφορετικά θα επανέλθουμε στην Ερευνητική Επιτροπή όπου εξακολουθούμε να έχουμε όλα μας τα δικαιώματα. Επίτροπε, είναι ασφαλώς ε, φυσιολογικό ενδεχομένως το γεγονός ότι σε κάποια κρατημέρια ασκούνται πρακτικές φοροαποφυγής και επιτρέπεται αυτή η φοροαποφυγή για το λόγο ότι πολύ απλά υπάρχει επιθυμία να προσελκύσουν μεγάλους ομίλους. Σε πρώτη, εκ πρώτης όψεως αυτό μπορεί να φαίνεται ως μια φυσιολογική λοιπόν πρακτική. Παρ' όλα αυτά, αυτή η φυσιολογική πρακτική περιλαμβάνει και ένα επικίνδυνο φάσμα δράσεων. Ως εκ τούτου, κύριε Γιούγκερ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε υπόψη σαν οποιαδήποτε μέτρα για την μείωση, τον περιορισμό των πρακτικών αυτών και για την αντιμετώπιση όσων σχεδιάζουν, προγραμματίζουν τέτοιους ε, κανόνες. Τα κράτη-μέλη, αναφέρθηκε, δεν απαντούν σε ό,τι αφορά τις ε, άδικες προλογικές πρακτικές. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι διτεθειμένα όλα τα κράτη-μέλη να προβούν σε σχετικέ δηλώσει και ότι κάποιοι ενδεχομένω να επιθυμούν να παραμείνουν προλαγική παράνταση. Αλλά μερικά από τα κράτη-μέλη αυτά έχουν προσχωρήσει σε πάρα πολλέ σημαντικέ συνθήκε και επτά εξ αυτών έχουν αγνοήσει τι υποχρεώσει αυτέ. Τι μέτρα λοιπόν χρειάζεται να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο τη ω θεματοφύλακα των συνθήκων και κατά συνέπεια να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των όσων προβλέπει η συνθήκη, αλλά και να διασφαλίσει πίστη προς ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Γιούνκερ, με προσοχή άκουσα τα όσα είπατε για έναν από τους επιτρόπους, ο οποίος ήταν υπεύθυνο που είναι υπεύθυνο για τον αναγωνισμό και διακόπτει δυστυχώς ο πρόεδρος, ο κύριος Μόνο. Μονό. Κύριε Μονό, είστε εδώ. Ο κύριο Μονό έχει το λόγο. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την παρουσία σα εδώ. Ξέρετε, πολλέ φορές οι χρονικές συγκυρίες είναι πολύ σκληρέ. Πριν από λίγα... Ε, εδώ, ε, πιο δίπλα, υιοθετήσατε ποσοστώσεις για τους μετανάστες. Εξ ονόματος ποιου το κάνετε αυτό ανθρωπισμός, αλληλεγγύη, όποτε σας βολεύει την χρησιμοποιείτε. Γιατί την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό την είχατε γραμμένη για 20 χρόνια όταν είχατε υιοθετήσει καταχρηστικές πρακτικές φορολογικές για να προσελκύσετε επιχειρήσεις στο Λουξεμβούργο, στη δική σας χώρα, αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού και αυτές είχαν ανέλθει στην ανώτερη διοικητική ιεραρχία της χώρας σας. Και σήμερα έρχεστε να μας μιλήσετε για το πώς ε, θα καταπολεμήσουμε ε, το optimization fiscal, την αναζήτηση δηλαδή του πιο προνομιούχου φορολογικού καθεστώτος ε, της εκάστοτε χώρας από πλευράς επιχειρήσεων. Όμως όταν ήσασταν Πρωθυπουργός, όταν ήσασταν Υπουργός, πότε πότε λάβατε την πολιτική απόφαση να να δουλέψετε υπέρ αυτού του ε, ευαγούσου σκοπού. Πάντοτε ε, παίρνατε αποφάσεις προς την αντίθετη ε, κατεύθυνση, οι οποίες ωφελούσαν μόνο τους επευθύνους των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν γίνεται ένας πρωθυπουργό μιας χώρας να μην ξέρει ότι η δική του φορολογική διοίκηση έχει συνάψει τέτοιου είδους φορολογικές συμφωνίες με, με ένα οικονομικό όφελος που βρίσκεται σε αστρονομικά επίπεδα. Είμαι πατριώτης και αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι οι Γάλλοι φορολογούμενοι υπέστησαν ένα τεράστιο βάρος γιατί ε, οι φόροι δεν συλλελέγησαν από επιχειρήσεις που πήγαν αλλού, όπου ευεργετήθηκαν. Νομίζω ότι για όλα αυτά μας οφείλεται πιο ειλικρινές απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Γιούγκερ και ο Επίτροπος Μοσκοβισή έχουν το λόγο για να απαντήσουν στην πρώτη σειρά των ε, ερωτήσεων. Παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Τουλάχιστον 20 ερωτήσεις ε, μου απευθύνθηκαν. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται στις απαντήσεις για να σας δώσω την δυνατότητα να μου πείτε αν δεν απάντησα. Προς τον κύριο Μπάλτ να πω ότι Τον άκουσα με φιλικό πνεύμα και όταν δήλωσε και ρώτησε τι θα απαντούσα στον ε, επιχειρηματία. Για μένα είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, σε κατά κανόνο ανταποκρίνονται και εκπληρώνουν τα φορολογικά τους κοντά. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να και πρέπει να φροντίσει για πιο πολύ δικαιοσύνη σε θέματα φορολογίας. Και αυτό έχει να κάνει και με το θέμα και της βάσης υπολογισμού. Θα πρέπει να το δούμε με νέο πνεύμα, με καινούργιο μάτι. Ελίζα Φερέρα. Σωστά υπέδειξε ότι προέκυψε αν και δεν μπορούσα να το ελέγξω στην πράξη, ότι αυτά που προέκυψαν από το LuxLeaks για μέσα των, του τύπου αποτελεί τελικά μια συνήθιση πρακτική για πολλά κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να το λέμε καν LuxLeaks ενδεχομένως το φαινόμενο, γιατί αυτό ενδεχομένως να μειώνει και να περιορίζει γεωγραφικά το ζήτημα και αυτό δεν ε, είναι παρά μια απόπειρα απλοποίησης. Ε, συμφωνώ με την κυρία με ζούμε στη ζούγκλα και θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια για τον ε, καθηγητή Λούκε και για το θέμα των Τη νομοθεσίας και του δικαίου για τι επιδοτήσει. Θεωρητικά έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Σχόλια εκτό μικροφώνου. Ναι, εσείς είστε καθηγητής. Εγώ έχω ασχοληθεί μάλλον με στην πράξη με το θέμα αυτό. Είναι διαφορετικό λίγο. Είναι διαφορετική η προοπτική. Είμαι, επίτροπος, ε, είμαι πρόεδρος Επιτροπής, αλλά αρνούμε να μπω στα νερά τη Επιτρόπου για θέματα ανταγωνισμού πιστεύω στην αυτονομία και την εξαρτησία των κινήσεων της Επιτρόπου και δεν πρόκειται να μπω στα πόδια της, αλλά συμφωνώ με σας, επειδή με ρωτήσατε ότι σε θέματα φορολογίας τίθεται θέμα κρατικής επιδότησης και πιστεύω λοιπόν ότι κάθε φορά που τίθεται το θέμα αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε και την πτυχή αυτή. Θα πρέπει και τα φορολογικά πλέον εκτίμεα να ελέγχονται κατά καιρό. Και αν υπάρχουν ε, ορθοί λόγοι για να υπάρχουν ε, αυτά τα αυτές τις ρυθμίσεις, ε, το εξετάζουμε. Κύριε Τόιρερ το κατά πόσον συναντήθηκα με επιχειρήσεις συμβουλευτικής. Όχι, ποτέ. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και από τους λίγους αυτή τη συνεδρίαση που δεν έχει συναντηθεί ποτέ με εκπροσώπους επιχειρήσεων συμβουλευτικής. Τους έχω παρακολουθήσει. Έχω παρακολουθήσει πώς ε, αυτές οι, αυτές οι εταιρείε ε, έχουν επαφές με διάφορους και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δεν θα αφήσω να μου πούνε τι θα κάνουμε στη φορολογική πολιτική εταιρείε οι οποίε άμεσα επηρεάζονται από αυτήν. Σα είπα ότι είχα αυτή την ε, είχα αντιμετωπίσει αυτή η φορολογική Επιτροπή με δίκαιο πνεύμα. Δεν ήμουν το υπέρ. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν υπέρ, ποιος ήταν κατά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κανείς δεν ήταν υπέρ τότε στις συναντήσεις του Συμβουλίου. Και το ποιος ήταν υπέρ νομίζω ότι το καταλαβαίνετε. Ένας μόνο ήταν υπέρ και ήμουν εγώ. Ε, μα το φτάνει όμως ένας. Αλλά καλό θα ήταν αν η πρόταση αυτή ε, θα έρθει να συμπεριληφθεί στην ε, έκθεσή σα. Νομίζω ότι ανταποκρίνεται πολύ στο πνεύμα των όσων έχει ω αντίληψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Λουξεμβούργο δεν ε, ε, άφησα να υπάρχει ένα καθεστώ φορολογικό ούτε το εφήβραφο, το φορολογικό καθεστώ φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, φορο απαλλαγής εις βάρον άλλων κρατών μελών. Υπερτιμάται και τις ικανότητές μου. Το Λουξεμβούργο είναι ένα κράτος δικαίου και η νομοθεσία προβλέπει ότι οι φορολογικές αρχές εφαρμόζουν το φορολογικό δίκαιο, όχι ο Υπουργός Οικονομικών. Το Λουξεμβούργο είναι μεγάλα του κάτω, αλλά μικρή χώρα. Και είναι μεγάλη ενεργία κατά των ε, παρεμβάσεων από τα Υπουργεία, ξέρετε. Αν υπήρχε τέτοια απόπειρα σε ένα τέτοιο μικρό μέρος όπως το Λουξεμβούργο, θα είχαν βγει στις εφημερίδες όλα αυτά μετά από δύο μέρες. Αλλά δεν έγινε γιατί δεν το έκανα ποτέ, γιατί ο επαγγελματισμός και η αποδοτικότητα της φορολογικής υπηρεσίας πράγματα ήταν γνωστή. Ρωτήσατε για την έκθεση Κρίκελ, κύριε Βουλευτά και Δεν ήξερα ότι τότε που έγινε η συνέντευξη του κυρίου Κρίκελ δεν περιλήφθηκε μία σελίδα. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτή η σελίδα. Ούτε τον ε, κάλεσα να την αφαιρέσει αυτή τη σελίδα γιατί δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η σελίδα. Αλλά φυσικά είναι το θέμα, ήταν θέμα πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν του ανέθεσα τη συγγραφή ενός άρθρου για την ε, φορολογική αποφυγή. Και τον τηλεφώνησα όταν έγινα υπουργό. Και του είπα ότι δεν ε, μου είπε ότι δεν μου ζήτησε η κυβέρνηση να αφαιρέσω εγώ τη σελίδα. Εγώ αποφάσισα να την αφαιρέσω. Γιατί δεν ε, ήταν κάτι που θεωρούσα απαραίτητο. Δήλωσε λοιπόν ότι αφαίρεσε τη σελίδα αυτή γιατί αυτή η έκθεση που είναι 216 πλην μία σελίδας δημοσιεύθηκε και επέκρινε για το tax ruling μια κυβέρνηση συγκεκριμένη και ήξερε ότι έχουμε σε θέματα φορολογίας 97 πρωτοβουλίες και εν πάση περιπτώσει έκρινε ότι έπρεπε να αφαιρεθεί, αλλά μπορείτε ασφαλώ να τα συζητήσετε και εσεί μαζί του. Εγώ συναντήθηκα με τράπεζες σε κάποιε περιπτώσει και με την Commerzbank συναντήθηκα. Αλλά είναι αρκετά φυσιολογικό αυτό. Όταν είναι κανεί πρωθυπουργό ή υπουργό οικονομία μια χώρα να συναντιέται και με τραπεζίτε σε κάποιε περιπτώσει, αλλά ποτέ με την Commerzbank δεν ε, Συζητήσα θέματα διαμόρφωσης του προλογικού του καθεστώτος. Η Commerzbank πάντα μου έλεγε τι φόρους ε, πληρώνει στο Λουξεμβούργο και πάντα παραπονιόταν. Και ε, εγώ πάντα έλεγα ότι οι τράπεζε που πληρώνουν φόρου στο Λουξεμβούργο να μην γνιάζουν να είναι γνώμονες που μπορούν να λειτουργούν και να πληρώνουν φόροι. Φόρους. και πολύ εδώ πέρα στην αίθουσα. Ξέρετε ότι δεν ήμουν από του αγαπημένου των ε, τραπεζών στο Λουξεμβούργο και σε ό,τι αφορά του whistleblowers, του πληροφοριοδότες, θα αναλάβουμε πρωτοβουλία ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί νομίζω ότι και το θέμα αυτό θα πρέπει να τύχει μια ευρωπαϊκή απάντηση. Κύριε Σβέν Κίγκολτ, ξέρετε, ξέρετε ότι δεν θα διαμόρφωνα το φορολογικό καθεστώ στο Λουξεμβούργο ποτέ έτσι ώστε να βλάψω άλλους ότι κανένα δεν, ήθελα, δεν μπορούσα να θέλω να βλάψω σκόπιμα. Στο θέμα της ε, εταιρικής και της ατομικής φορολογίας ήθελα να βοηθήσω για παράδειγμα το Βέλγιο βάσει μια συμφωνίας ε, μεταξύ του Βελγίου και της ε, Λουξεμβούργου ε, ε, παίρνει 600 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος για, από, τους, από τα άτομα που εργάζονται κοντά στα σύνορα και περνάνε τα σύνορα για να δουλέψουν και σε ό,τι αφορά τα θέματα αλληλεγγύης με τους γείτονες Νομίζω ότι πολλά μπορώ να σας πω ως παραδείγματα και προς τις δύο πλευρές. Ο πρόεδρος ε, Πάκας και ο κύριος Γκίγκολτ έθεσαν ένα ερώτημα το οποίο ενδεχομένως να πρέπει να απαντήσει ο Επίτροπος Μόσκοβίση, ο κύριος Μονό. Ναι, συγγνώμη, λέει ο κύριος Γκίγκολτ, αλλά αυτό δεν αποτελεί καμία απάντηση στο ερώτημά μου για την πρόσβαση στα δημοσία έγγραφα. Ναι, δεν καταλαβαίνω αυτή τη βιασύνη. Σα είπα, μπορείτε να ακούσετε και φαντάζομαι να είπα ότι θέλω να θα απαντήσει ο κύριο Μουσκαπησί. Όχι, θέλω από εσά, κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή γιατί δικιά σα ευθύνη είναι. Όχι, λέει ο κύριο Γιούνκερ, σήμερα δικαίω επισημάνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, ε, ανέλαβε για την προώθηση του, των εγγραφών αυτών. Ο κύριος Μοσκοβισή θα απαντήσει θα απαντήσει στην ερώτηση και δεν είστε καθόλου αρμόδιοι να αποφασίσετε ποιο θα πρέπει να το απαντήσει αυτό από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιο είναι σε θέση να απαντήσει σωστά την ερώτηση αυτή. Δεν ε, θέλω να σας απαντήσω γιατί με διακόπτουν συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει αναφέρεται το όνομα του κυρίου Μάριου Σκόλ, τον οποίο είχα συναντήσει ως Υπουργό Οικονομικών εγώ και εκείνος προϊστάμενος στη φορολογική διοίκηση, αλλά δεν είχα ιδιαίτερες σχέσεις μαζί του. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δώσει καμία εντολή ούτε διαταγή στη Λουξεμβούργια φορολογική διοίκηση. Δεν είναι δική μας αντίληψη αυτή για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Δεν παρεμβαίνει πολιτική εξουσία στη διοίκηση, τη φορολογική. Περσεβεράρε μου. Όταν εσεί το λέτε αυτό σίγουρα θα ξέρετε γιατί μιλάτε. Ο επίτροπο Μοσκοβισή παρακαλώ. Ναι, δύο λόγια θα ήθελα να πω ε, για δύο θέματα. Ένα ουσίας και ένα επί τη διαδικασίας ε, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σα. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριο Μπάλτσα, Πάσκα και Τόιρε, η κυρία αυτή οι συνθήκες του ανταγωνισμού, στρεβλού ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων από τη μία και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την άλλη. Αυτό είναι το πρόβλημα και αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν φορολογικό βάρος μεγαλύτερο κατά 30% πολύ συχνά έναντι των μεγάλων ομίλων και δεν έχουν και το σύνολο των πληροφοριών στη διάθεσή τους. Θα πρέπει να ασκήσουν αυτές πίεσεις στα Συμβούλια Υπουργών έτσι ώστε να έχουμε ένα κοινό ε, παρονο, παρονομαστεί. Να δουλέψουμε περισσότερο και για το CCCTB και για ε, το ε, την καταπολέμηση των προνομιακών φορολογικών καθεστώτων, αλλά και για την ενοποιημένη κοινή βάση για φορολόγηση εταιριών. Και θα πρέπει να διοργανώσουμε μια κατάσταση στην οποία από τη μία να μην υπάρχουν ε, εξαιρετικά αδύναμες φορολογήσεις και ε, να μην, είναι, να μην επιτρεπτό πλέον να μην έχουν πρόσβαση σε ε, τέτοιου είδους καθεστώτα μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί είναι σε κατάσταση μειονεκτήματος στρατηγικού και ανταγωνιστικού. Από εκεί και πέρα για το θέμα της διαδικασίας του αιτήματο ε, πληροφόρησης που υποβάλλεται σε μένα, γιατί εγώ είμαι αρμόδιος επίτροπος με το σχετικό χαρτοφελάκιο. Στις 31 Αυγούστου σας έδωσα μια πρώτη απάντηση η οποία δεν σας ικανοποιεί πλήρως. Το κατάλαβα γιατί συζήτησα με τον κύριο Λαμασούχ. Θα επανέλθω. Ποτέ δεν αρνήθηκα να διαβιβάσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα έγγραφα που είχα στη διάθεσή μου. Ωστόσο υπάρχει ένα όριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει την εξουσιοδότηση να διαβιβάσει ορισμένα έγγραφα χωρίς την έγκριση των κρατών μελών. Είναι κανόνες εμπιστευτικότητας που προκύπτουν από την ε, συμφωνία, ε, τη ε, σύμβαση και προβλέπετε κάτι τέτοιο ρητά. Γνωρίζω ότι η απάντηση δεν σας ικανοποιεί και ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις. Συμφωνώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώθηκε ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι κατά της δυνατότητας να μοιραστούν τα κράτη-μέλη έγγραφα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά επιθυμούν τα κράτη-μέλη να τηρηθούν οι κανόνες εμπιστευτικότητας. Εκεί λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε, αυτό πρέπει να εξισορροπήσουμε για μένα είναι επιτακτική ανάγκη το Κοινοβούλιο να ασκήσει το δικαίωμα πληροφόρησή του και από την άλλη διαδιατηρηθεί το σύστημα τη εμπιστευτικότητα που επιζητούν τα κράτη-μέλη. Άρα να ζητούμε πρακτικού τρόπου εφαρμογή, λεπτομέρειε εφαρμογή του πώ θα συγκεράσουμε αυτά τα δύο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη μαζί με εσά να θεσπίσουμε ένα πλαίσιο για την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούν να εξουσιοδοτηθούν άτομα να λάβουν γνώση των εγγράφων και θα πρέπει η πρόσβαση να δίδεται σε κάθε πολιτική ομάδα. Τα κράτη-μέλη ε, ήρθαμε σε επικοινωνία με αυτά, εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας είπαν ότι μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και σε ρύθμιση εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή και να το δούμε το θέμα για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, ωστόσο να τηρηθεί το δικαίωμα της πρόσβασης των εγγράφων διατηρώντας πάντοτε την εμπιστευτικότητα. Δηλαδή βρίσκουμε το σωστό μείγμα πολιτικής έτσι ώστε να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα και οι πολιτικές ομάδες από την άλλη να έχουν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα. Γίνεται προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ ο πρόεδρος Λαμασούχ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε επίτροπε. Έχουμε ένα πρόβλημα χρονικό, ένα πρόβλημα χρόνο. Ε, σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μείνατε 15 λεπτά παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη άλλωστε το γεγονός ότι καθυστερήσαμε γιατί έπρεπε να πάμε στην Ολομέλεια να ψηφίσουμε. Ωστόσο έχουμε 8 ομιλητές που θα υποβάλουν ερωτήσεις και αν θέλουμε ο Πρόεδρος και ο Επίτροπος να μας απαντήσουν, προτείνω ο κάθε ομιλητής, ο κάθε ερωτών να μην ξεπεράσει το ένα λεπτό. Μία ερώτηση για ένα λεπτό. Η κυρία Ντανούτα Χιούμπνερ, εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Αλέν. Θα ήθελα να αφυπνίσω την πολιτική διέστηση του Πρόεδρου Γιούνκερ και να σας ρωτήσω, πιστεύετε πραγματικά ότι μπορούμε να πετύχουμε την κανονικοποίηση των προνομιακών φορολογικών καθεστώτων μέσω της διαδικασίας του benchmarking και ενθαρρύνοντας τα κράτη-μέλη να τα περιλάμβουν στην εθνική τους νομοθεσία ή θα πρέπει να νομοθετήσουμε έτσι ώστε το πρόβλημα να ρυθμιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα το πακέτο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκεί θα βοηθούσε αν είχαμε μία, έναν αρνητικό ευρωπαϊκό κατάλογο θεμάτων που δεν θα πρέπει να μπει στα tax ruling, στα ειδικά φορολογιακά καθεστώτα, αλλά θα πρέπει να μπει στο κανονικό φορολογικό καθεστώς της κάθε χώρας. Ο Πίτερ Ζήμεν για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από επισκέψεις σε πολλά κράτη-μέλη και εξέταση διάφορων ε, γράφων διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολύ αμφισβητής ενώ το θέμα της φορολόγησης ε, των μεγάλων ε, ομίλων μπορεί να είναι νόμιμη αλλά να, ενδεχομένως να εμπίπτει και στο καθεστώς για τις επιδοτήσεις, για τις κρατικές βοήθειες και σε μεγάλο ποσοστό αυτό αναφέρεται ως κανονικό καθεστώς. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφάνεια αν θέλουμε να προσεγγίσουμε την κατάσταση και χαίρομαι που ο κύριος Μοσκοβίση μίλησε και ανέφερε ότι θα μας χορηγηθούν τα έγγραφα αυτά προκειμένου και το απόρριτο να τηρήσει και να έχει πρόσβαση. Δεν θα αποδεχτούμε όμως από τα κράτη-μέλη, δεν θα αποδεχτούμε να μην μας διαθεθούν έγγραφα το Κοινοβούλιο διατηρεί την, ε, το απορριτό και τον τρόπο μπορούμε να τον βρούμε. Αλλά το να δώσουμε όχι ως απάντηση είναι απαράδεκτο, διακόπτει ο Πρόεδρος. Δυστυχώς, δυστυχώς, ε, αγαπητέ συνάδελφε. Για το ΕΛΚ, ο Παύλο Θέλβα. Παύλο Θέλβα για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αναμφίβολα το Lux Leaks είναι η απόδειξη του ότι χρειαζόμαστε μια φορολογική Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και ευκαιρία να τη δηλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Να μην χάσουμε την χρονική συγκυρία Επίτροπε Μοσκοβισή και ο κύριος Βάλς, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, το είπε ότι ένα από τα προβλήματα της Ευρώπης είναι η αντιαγωνιστικότητα και κυρίως η ανταγωνιστικότητα των μικρομεσών επιχειρήσεων πλήττεται τα μάλα και αυτές είναι που δημιουργούν απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν πρέπει να θέτουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μη ανταγωνιστική και μειονεκτική θέση. Χαίρομαι γι' αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής. Δεν αρκεί όμως. Χαίρομαι και χαιρετίζω αυτά που, για αυτά που, παρατηρήσα, που παρουσιάσατε σήμερα εδώ, όμως δεν αρκεί ούτε αυτό. Πρέπει να τα εφαρμόσετε, Επίτροπε Μοσκοβισή, το συντομότερο δυνατό και να τηρήσετε τις δεσμεύσει σας. Να υποσχεθείτε ότι άπαξ και εφαρμοστεί, ε, τότε δεν θα ξαναπροκύψει και δεν θα ξαναζήσουμε αυτό που ζήσαμε πρόσφατα με το Λάξλεξ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ, Αναλύ Ντότς. Ευχαριστώ. Σύντομα και άμεσα, ε, συγγνώμη, καταρχήν έχουμε την απώλεια του μηχανισμού, αυτόματου μηχανισμού μετά την CCCTB ε, και πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο μηχανισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί για επιθετική φορολογική ε, πολιτική ε, ε, μπορεί λόγω αυτού του μηχανισμού να αυληθεί το αποτέλεσμα της CCCTB. Και έπειτα τι θα κάνετε με τους φορολογικούς παραδείσους και έπειτα μπορείτε και οι δύο να παραπέμψετε την ανάγκη οι μη πολυεθνικές και οι μη, και ιδιαίτερα να ληφθούν υπόψη όταν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα από τις διαβουλεύσεις για την CBCD. Ευχαριστώ αγαπητή Αναλύζη. Είστε Λάγκη. Κοιτάξτε, τους τύπου θα τους αφήσω. Ε, σας ευχαριστώ που ε, είστε εδώ, αλλά η ερώτησή μου είναι ε, πολύ κέρια. Είπατε ότι μπορείτε Ε, δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε εκθέσεις όταν τα κρατη μέλη αντιτίθεται στην δημοσίευσή τους. Το 1999 υπήρξε μια έκθεση για τις διοικητικές πρακτικές στα κρατημέλη. Νομίζω πως είναι πολύ σωστό να γνωρίζουμε, όχι μόνο για το tax rulings, αλλά για την ποικιλία των διοικητικών πρακτικών. Έγινε από τη Siemens και η Siemens με από, μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τότε δεν δημοσιεύθηκε γιατί υπήρχαν προβλήματα στο Συμβούλιο. Νομίζω πως κύριε Μοσχοβίτη, ε, τότε ήσασταν εσείς στο Συμβούλιο ως Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας. Μπορείτε να μας πείτε από την εμπειρία σας ποιο ήταν το πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσαμε να δημοσιεύσουμε, η Κομισιόν δεν μπορούσε να δημοσιεύσει την, ε, την έκθεση Siemens ε, και επειδή υπήρξε ενημέρωση για το 2009 και σχετική έκθεση για τα νέα κράτη-μέλη. Μπορούμε να το έχουμε και αυτό. Ενημερωμένο και πλήρη την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, ήταν σαφή η ερώτησή σας. Ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Μα ζητήσατε Είπατε ότι θα μας βοηθήσετε, αλλά η προϋπόθεση της πρόσβασης στα εγγραφά θα πρέπει να είναι καλύτερη από ό,τι τώρα. Για τα αναχώρα, αναχώρα εκθέσεις, ξέρετε ότι το κοινοβούλιο μας είναι πολύ επιθετικό. Και καταλαβαίνουμε ότι στο Συμβούλιο υπήρξε ε, απροθυμίες για τη δημοσίευση των εκθέσεων από τον ε, των εκθέσεων αναχώρα. Μα πώς γίνεται αυτό κάναμε αναχώρα για τις πολυεθνικές, για τις τράπεζες, μα είναι δημόσια. Γιατί στο καλό υπάρχει πρόβλημα για αυτή την υπόθεση. Ε, και αυτά τα θέματα δίθεν για τον ανταγωνισμό δεν μας πείθουν. Γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα της ψηφιακής οικονομίας δεν θα λυθεί παρά μόνο μία, μέσω μιας οριζόντιας φορολόγησης. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε την CCTB, την Ενωπημένη Κοινή Βάση για τη Φορολόγηση των Εταιριών και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν διαφορετικά να καλύψουν αυτή τη φορολογική βάση που διαφεύγει ε, της φορολόγησης. Εσείς λοιπόν υπέρ των τεσσάρων σε, σε, Κύριε Νίτερμαϊερ, σας ευχαριστώ πάρα πολλά. Καταρχά, για ό,τι αφορά το CCTV, ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντυπωσιακό πρόγραμμα για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης υπέρ τη δικαιοσύνη στη φορολογία, υπέρ των επιχειρήσεων. Να ρωτήσω λοιπόν, πώ σκοπεύετε να πείσετε τα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν το CCCDB σε ό,τι αφορά ε, του φορολογικού φορολογικούς Δεν ε, είμαστε βέβαιοι για την έκταση του προβλήματο και δεδομένης ε, της χαμηλής απόδοσης φορολογικών εσόδων Τη απόδοση των φορολογικών εσόδων δεν είναι το βασικό μα πρόβλημα, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα των BEPS σε ό,τι αφορά τη διάβρωση της βάσης και τη μεταφορά των κερδών, σε ό,τι αφορά τα... Το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κομφεράτη. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα εκ νέου να επιστήσω την προσοχή σας στις εκθέσεις, εκθέσεις ανά χώρα. Το ε, προηγούμενο Ιούλιο το Κοινοβούλιο έκανε ένα κείμενο που σχετίζεται με το θέμα της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων που τροποποιούσε την οδηγία accounting. Για τους μετόχους είναι πολύ σημαντικό να έχουν αυτές τις πληροφορίες για να μπορούν να αποφασίσουν πώς θα επενδύσουν αλλά και για να υπερασπιστούν τη φήμη τους. Ε, Το θέμα της εκτίμησης αντικτύπου έχει λυθεί. Όταν ψηφίστηκαν οι κανόνες σε σχέση με τα δημοσιονομικά Ινστιτούτα, έγινε η σχετική ψηφορία και ήταν θετική έκβαση. Αν θέλετε διαφάνεια, υπάρχει μια κοντινή ευκαιρία και είναι σημαντική. Θα ξεκινήσουν τριμερεί στι επόμενε μέρε. Υπάρχει μια ανεξήγητη εχθρότητα από πλευρά των κατών μελών, αλλά είναι καλή ευκαιρία για να εισαχθεί αυτή η καινοτομία που εξυπηρετεί ε, ακριβώς ε, μετά ένα χρόνο από το LuxLeaks. Όταν τέτοιου είδου ε, διατάξει δεν, δεν είχαν ακόμα εγκριθεί από τα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ συνάδελφοι για την αυτοσυγκράτησή σα σε αυτό το τόσο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Εν μεταξύ έχουμε πλέον την παρουσία τη Επιτρόπου και Μάργαρετ Φερσχάγκερ, την οποία χαιρετίζω. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Και κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, παρακαλώ να απαντήσετε χωρίς να πάρετε πάρα πολύ χρόνο από την επόμενη ακρόαση. αλλά είμαι βέβαιος ότι μαζί με την Επίτροπο Αρμόδια του Ανταγωνισμού θα βρείτε κάποια συνεννόηση. Το θέμα των ε, ε, μεταβιβάσεων των φορολογικών θα το αφήσω στην κυρία Φεστάγκερ, το γνωρίζει καλύτερα και για τα λοιπά θα δώσω το λόγο στον κύριο Μοσκοβισή. Θα παραμείνω για να παρακολουθήσω τη συζήτηση για λίγο. Όμως έχω να συναντήσω και πολλούς υπουργούς Θέλω να σημειώσω ότι είμαι πάντοτε δίπλα στον Πιέρ Μοσκοβισή, όποτε με χρειαστεί, είμαι στη διάθεσή σας. Το φαινόμενο που εσείς προσπαθείτε να περιγράψετε ως lax leaks είναι πολύ πιο ευρύ και ίσως το πρώτο συνθετικό της λέξης αυτής θα πρέπει να αλλάξει και να περιλάβει πολύ περισσότερες έννοιες. Ευχαριστώ πολύ. Bien. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Πέντε ομάδες ερωτήσεων σημείωσα. Πρώτον, για τα προδομιακά φορολογικά καθεστώτα. Πράγματι δεν είναι μια πρακτική που ακολουθείται μόνο στο Λουξεμβούργο και εγώ ήμουν Υπουργό Οικονομικών σε άλλη χώρα και είναι αληθές ότι δεν είναι κακό να μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να προβλέψουν τον εταιρικό φόρο που θα καταβάλουν. Αυτό το οποίο καταδικάζουμε είναι η σκοτεινότητα, η σκοτεινιά το ότι όλα αυτά είναι κρυμμένα και κρυφά και δεν τα γνωρίζουν όλοι όπως πρέπει παρά μόνο ορισμένε πολιεθνικέ οι οποίε τα αξιοποιούν για να ε, κερδίσουν σε βάρο τη μία ή τη άλλη χώρα. Και γι' αυτό στι 6 Οκτωβρίου στο Συμβούλιο Κοφίν ελπίζω ότι η πρότασή μα θα τύχει έγκρισης και θα εφαρμοστεί από τι αρχέ του 2016. Ελπίζω η πρόοδο επί της διαφάνειας να συνοδευτεί από ε, περαιτέρω δράσεις από τα κράτη-μέλη ούτως ώστε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια και να μην ε, δημιουργείται μια κατάσταση κατά την οποία η μία χώρα επιβαρύνει μια άλλη ουσιαστικά. Τώρα, ως προς το άξι, στην ενοποιημένη κοινή φορολογική βάση για τη φορολόγηση των εταιριών. Είναι ένα καλό σχέδιο αυτό. Όταν όμως είναι κανείς επίτροπος πρέπει να παντρέψει την προσέγγιση του εφικτού με την προσέγγιση του ε, ε, πιθανού, του εφικτού με του επιθυμητού μάλλον και γι' αυτό υθετήσαμε την προσέγγιση ανά δύο στάδια. Το γεγονός ότι ξεκινούμε από την επίτευξη κοινής φορολογικής βάσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι παρετούμαστε από την ενοποίηση και όλας αυτής. Αλλά τώρα ασχολούμαστε με την δημιουργία κοινή φορολογική βάσης γιατί θα ήταν προθύστερο ε, να ενοποιήσουμε ανώμια πράγματα. Το ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση δεν σημαίνει ότι βάζουμε τη δεύτερη που είναι και η πιο σημαντική στο σιρτάρι και στο χρονοτούλαπο. Η δική μου ε, θέση είναι ξεκάθαρη. Είχαμε δημόσια διαβούλευση, είχαμε αξιολόγηση αντικτύπου, όχι για να ξεδοδιάσουμε το reporting αναχώρα, αλλά για να δούμε πώς μπορούμε να το υλοποιήσουμε από τη μία χωρίς να βλάψουμε τις επιχειρήσεις από την άλλη. Και με βάση τη δημόσια διαβούλευση θα πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Σε κάθε περίπτωση δεν το κάναμε για να ξεφύγουμε από το θέμα και να ε, το αποφύγουμε. Ο κύριος Χίλ ασχολήθηκε με αυτό γιατί ήταν στο χαρτοφυλάκιό του, επίτροπος. Τώρα το θέμα έρχεται στα δικά μου χέρια. Στη δική μου αρμοδιότητα θα συνεργαστώ με τον πρόεδρο της Επιτροπής, με όλους εσάς, έτσι ώστε να έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση μέχρι τις αρχές του 2016. Τέταρτο ερώτημα, πρόσβαση στα έγγραφα. Και όπως το είπα και προηγουμένως, και σας νιώθω βαθύτατα, σας εξήγησα το θέμα της εμπιστευτικότητας Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για να υπάρχει σωστή ισορροπία μεταξύ της δικής σας απέτησης για διαφάνεια, την οποία καταναώ πλήρως, και το αίτημα των κρατών μελών για εμπιστευτικότητα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να έχει κεντρικό ρόλο στο μηχανισμό για τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα, τα tax rulings, και θα πρέπει όλοι αυτοί οι κανόνες και προϋποθέσεις να ισχύουν και για την ίδια. Έχω το, την έκθεση Simon Simon του 1997. Ήταν μια έκθεση που είχε εγκριθεί στο Συμβούλιο Γενικών Επιπροθέσεων. Τότε δεν είχαμε εκοφήν ούτε ανταγωνιστικότητα Συμβούλιου. Ο Αλέν Λαμασούχ κάτι θα ξέρει γιατί ήταν προκάτοχός μου. Και ε, ήδη βλέπετε τι πολλή δουλειά έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τότε μέχρι σήμερα. Τώρα, ως προς το ΦΠΑ, Πιστεύουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2016 θα έχουμε ένα οριστικό καθεστώς για το θέμα αυτό. Και ολοκληρώνω για να μην μακρηγορώ κιόλα λέγοντας ότι στο ερώτημα ποια είναι η βούληση και ο κινητήριος μοχλός πίσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώ λέγοντας ότι εμείς δρούμε ε, υπό την πίεση των πολιτών που πραγματικά πιστεύουν ότι το θέμα είναι επίγον και εσείς ε, διερμηνεύετε αν τα λόγια των πολιτών οι οποίοι δεν θέλουν πια ε, να υπάρχει ε, συγκάλυψη και να είναι, γίνονται όλα αυτά κρυφά. Και είναι πράγματα για τα οποία αντιλαμβάνομαι, κατανοώ και συμφωνώ πλήρως. Θεωρώ ότι η παρουσία σας είναι ατού και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε εδώ για να περάσουμε το μήνυμα των Ευρωπαίων πολιτών και να ξεμπλοκάρουμε ε, διαδικασίες ε, έναντι αυτών οι οποίοι είναι πιο επιφυλακτικοί και οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν με πιο αργά ε, βήματα και καθόλου δεν τους μέμφωμε και καθόλου δεν τους υποπτεύουμε. Απλά μερικές φορές οι διαδικασίες είναι δίσκαμπτες, από την άλλη οι πολίτες επίγονται και θα πρέπει να έχουμε μια επανάσταση διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και διαφάνειας ε, αποτελεσματικότητας ε, και ε, σωστής λειτουργίας. Αυτά τα δύο, όλα αυτά μπορούν να συνδυαστούν. Ένα σύστημα που είναι πιο διαφανές θα είναι και πιο δίκαιο και πιο αποτελεσματικό. Και έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι θα είναι πρωτοπόρος σε ένα διεθνές κίνημα το οποίο την ξεπερνά άλλωστε. Αυτή ε, είναι η αποστολή μου, αυτή την αποστολή μου έχουν αναθέσει και χαίρομαι διότι θα την υπηρετήσω και θα έρχομαι συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα συζητούμε όλα αυτά και να στηρίζομαι πάνω σας. Θεωρώ ότι η δική σας επιδητική επιτροπή είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στήριξης εμού και της προσπάθειάς μου. Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, και εμείς θα κάνουμε το παν για να έχουμε όσο δυνατό μεγαλύτερη και καλύτερη πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες. Θα συνεργαστούμε μαζί σας Επιμένω σε κάτι που αναφέρθηκε σε μια πρόσφατη συνάντησή μας. Ως προς την ενοποιημένη κοινή φορολογική βάση για τη φορολογήση των εταιριών, για να κερδίσουμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε, καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει τροπολογίες στο σχέδιο κειμένου που έχει τεθεί επιτάπητος πριν από τρία χρόνια. Καλύτερο αυτό παρά να ξεκινήσει από το μηδέν είναι πιο σημαντικό για να διατηρούμε την πίεση που ασκούμε στις κυβερνήσεις και να τις υποχρεώνουμε να πάρουν αποφάσεις τάχιστα. Για να το καταφέρουμε πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε μια γρήγορη και ταχεία διαδικασία. Μπορούμε λοιπόν τώρα να αποδεσμεύσουμε τον Επίτροπο Μοσκοβισή και να καλέσουμε την Επίτροπο Φεστάγκερ να πάρει τη θέση του. Και συνεχίζουμε ευθύ αμέσως. So, I Μάλιστα. Να προτείνω λοιπόν να ξαναξεκινήσουμε. Ε, θα κάνω κάποιε αγωγικέ παρατηρήσει και μετά ο πρόεδρο Γουαλτιέρη θα εξασφαλίσει και την προεδρία μέχρι το τέλο τη ε, συνεδρίαση. Να ευχαριστήσω την Επίτροπο ε, για τον ανταγωνισμό. Καταρχήν για την πνεύμα συνεργασία που τη διακρίνει από την πρώτη μέρα για τι εργασίε τη Επιτροπή Τάξη και Έκονα, για την καταπολέμηση τους ε, φορολογικής, ε, του, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ως εθνικού μέσου. Απαντήσατε στο ερωτηματολόγιο μας ήταν αρκετά λεπτομερές μέσα στο πλαίσιο των πληροφοριών που μπορείτε να μας δώσετε γιατί ξέρουμε ότι στον ανταγωνισμό έχουμε πολύ συγκεκριμένους κανόνες είναι πολύ σημαντικό όμως για μας στη φάση όπου εργαζόμαστε για το σχέδιο έκθεσης και πριν να εγκρίνουμε την τελική έκθεση στην Επιτροπή και μετά στην Ολομέλεια να έχουμε τη δική σας αίσθηση, την δική σας άποψη για τα ερωτήματα που θα σας τεθούν από τους συναδέλφους και όσον αφορά τα διδάγματα που αποκομίζετε από τις έρευνες που εσείς ξεκινήσατε ή που συνεχίζετε μετά από ε, αφού έχουν ξεκινήσει από διάφορους προκατώ, από τον προκάτοχό σας. Ε, ευχαριστώ και σας δίνω το... και δίνω μάλλον την προεδρία στον πρόεδρο Γουαλτιέρη. Ευχαριστώ Αλέν. Να σας ευχαριστήσω και εγώ για την οργάνωση αυτής της κοινής συνεδρίασης να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Φερστάγκερ με την οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Και στην ετησία έκθεση πρωτοβουλία ε, για τον ανταγωνισμό. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή. Η κυρία Λάγκερ, ο Βέρνερ Λάγκερ θα το παρουσιάσει τον Οκτώβριο. Και ξέρω ότι τελευταία σε εμφάνιση στην ΕΚΟΝ 14 Ιουλίου ήταν στις 14 Ιουλίου και χρειάζεστε πιο πολύ χρόνο για τις ε, έρευνες ε, κατά των κρατών μελών σε θέματα χρήματα οικονομικά και από την άλλη πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη τακτικής ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά το, την κατάσταση και το πώς πάνε τα πράγματα. Άρα θεωρώ ότι αυτή η συνάντηση είναι εξαιρετική ευκαιρία για να το πράξουμε αυτό. Να δώσω το λόγο λοιπόν στην Επίτροπο και μετά θα ακολουθήσει ο γύρος ερωτοπαντήσεων. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και για την πρόταση. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην κοινή συνεδρία της Επιτροπής Τάξη και Εικόν. Καταρχάς, να σας συγχαρώ για το έργο των εισηγητών κύριε Βρέιρα και Μάικλ Τόιρερ για το σχέδιο έκθεσης για την έκθεση της Επιτροπής ε, Τάξη και την κυρία Τότς και τον κύριο Λιντεμάιερ για την δική τους δουλειά σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο follow-up από την πλευρά της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Το τονίζω αυτό ότι οι συγκεκριμένες θέσεις και οι συγκεκριμένες προτάσεις και η ένταση της εργασίας είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα προκειμένου να διατηρηθεί η κεκτημένη ταχύτητα. Η ορμή είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για το σχέδιο εκθεσής ότι έχει γίνει μια σωστή και εντελεχή ανάλυση. Ε, περιλαμβάνονται συστάσεις σε μεγάλο εύρος τομέων και πραγματικά είναι συνεκτικότητη Το σχέδιο έκθεσης επίσης επισημαίνει και αφιερώνει προσοχή στο θέμα του κρατικού του ελέγχου των κρατικών βοηθειών επενδύσεων και ορίζω το γεγονός ότι επισημαίνεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο το στοιχείο αυτό για να υπάρχει πιο δίκαιο ανταγωνισμό, πιο δίκαια αφορολογία στην Ευρώπη. Έχουμε κοινό στόχο, ξέρετε, και μάλιστα είναι φιλόδοξο ο στόχο αυτό. Θα πρέπει σκληρά να εργαστούμε για να τον πετύχουμε. Θέλουμε να υπάρχει δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των ε, πολυεθνικών και των μικρομεσαίων. Ω επιτοπλίστων, εκεί εστιάζεται το θέμα. Μπορεί να υπάρχει φυσικά ανταγωνισμός, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν ακολουθούν τους ίδιου φορολογικού συντελεστές τα ίδια φορολογικά προγράμματα. Θα ήθελα περαιτέρω να επισημάνω εδώ σήμερα το ότι η ότι ο έλεγχος των κρατικών επιδοτήσεων μπορεί πραγματικά να πετύχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά. αλλά ότι επίσης θα πρέπει να συμπληρωθεί και από άλλα εργαλεία αν θέλουμε όντως να πετύχουμε ε, συνεκτική φορολόγηση στην Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων. Μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι καμία εταιρεία δεν θα λαμβάνει πλέον εξήματα δικαιολόγητα. ότι δεν υπάρχει προνομιακή μεταχείριση και επιλογή κάποιων. Με άλλα λόγια, ότι όλες οι εταιρείες της χώρας θα τη χάνουν ίσες αντιμετώπιση. Είτε είναι μεγάλε, είτε είναι μικρέ στο είτε προέρχονται από τον χύψη κλάδο και με οποιαδήποτε τύπο ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να πετύχω όταν θέτουμε του στόχους για την κρατική για τις κρατικές επιδοτήσεις. Οι αποφάσεις σε αυτές τις περιπτώσεις ελπίζω να θέσουν σημαντική, σημαντικό προηγούμενο σε ό,τι αφορά τον τομέα των κρατικών επιδοτήσεων. Εγώ δεσμεύομαι σαφώς να χρησιμοποιήσω το εργαλείο αυτό κατά οποιοδήποτε ευρωλογικού μέτρου που στρεβλώνει σοβαρά τον ανταγωνισμό και φυσικά θα διστάσω να αναλάβω και την ε, δράση που χρειάζεται όταν για παράδειγμα μια επιχείρηση Κρίθεί ότι έχει πλέον εκτίματα τα οποία στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και τα οποία δεν πρέπει να υπάρχουν. Αλλά ο έλεγχο των κρατικών επιδοτήσεων, ξέρετε, έχει και, και αυτό στα όρια του. Αυτά τα όρια τα ορίζουν οι συνθήκε. Είναι σαφέ ότι δεν μπορούμε να επιλύσουμε τα πάντα με το εργαλείο αυτό παρά το γεγονό. Ε, έχουμε λοιπόν το σπυρί στο χέρι, δεν μπορούμε να χτυπήσουμε όλα τα καρφιά και δεν είναι όλα καρφιά. Χρειαζόμαστε και πιο γενικά μέτρα συγκεκριμένα για να κλείσουμε τα παραθυράκια, για να εγγυηθούμε μεγαλύτερη διαφάνεια, πολύ περισσότερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά την εταιρική φορολόγηση. Και γι' αυτό λοιπόν η συζήτηση που κάνατε με τον ε, πρόεδρο Γιούγκερ και τον Επιτροπό Μοσκοβισή είναι τόσο σημαντική. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε χωρί τέτοιε συζητήσει. Ε, βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε ποιε είναι. Ποιοι είναι οι περιορισμοί του ελέγχου των κρατικών επιδοτήσεων σε ό,τι αφορά την επιστροφή πόρων ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αντιμετωπίζει το εργαλείο αυτό τη στρέβλωση των ανταγωνισμού, μεταξύ των εταιριών. Αν ανταγωνισμός είναι ήδη στρεβλός. Το σωστό είναι να επιδιορθωθεί η κατάσταση σε σχέση με το πριν την περίοδο χορήγηση τη επιδότηση. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενο θα πρέπει να πάρει τα χρήματα του πίσω ή τουλάχιστον να επιστραφούν στον κρατικό προπολογισμό προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για κάποιο νόμιμο σκοπό. Και αυτή η επιστροφή λοιπόν των ε, επιδοτήσεων είναι ένα νόμιμο μέτρο το οποίο ακολουθεί τους εθνικούς κανόνες και τα κρατημέλη μπορούν ασφαλώς να επιλέξουν την διαδικασία αρκεί να επιτρέπεται η άμεση και αποτελεσματική επιβολή της απόφασης επιστροφής που έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα τώρα να σας αναφέρω τα όσα είχαμε συζητήσει και το Μάιο για να σας πω που βρισκόμαστε. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τι πρακτικέ tax ruling για τα ειδικά προνομιακά φορολογικά καθεστώτα των κρατών μελών. Θα θυμάστε ότι τον Μάιο η συνεργασία με τις, ε, η συνεργασία των κρατών μελών για την μελέτη ανά κράτος μέλος δεν ήταν ακόμα ιδανική. Κάναμε λοιπόν μια συλλογή συνθήκων και Ζήτησα λοιπόν από τις υπηρεσίες μας να συλλέξουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονταν ε, για να μπορέσουμε να λάβουμε αποφάσεις. Και με χαρά μου μπορώ να σας ανακοινώσω ότι πλέον όλα τα κρατημέλη συνεργάζονται με τις έρευνες αυτές. Μετά από την έκδοση δικαστικών εντολών, λοιπόν, συλλέχτηκαν τα στοιχεία αυτά. Συλλέξαμε λοιπόν ένα μεγάλο αριθμό περαιτέρω tax rulings και σε άλλα κράτη-μέλη προκειμένου να αναλύσουμε αυτά τα φορολογικά καθεστώτα και στην παρούσα φάση, παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίε μου εξακολουθούν να αναλύουν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι η διαδικασία για τη χορήγηση τέτοιων προνομιακών φορολογικών καθεστώτων συνάδει ουσιαστικά με τα όσα προβλέπει ο Υπάρχουν λοιπόν και καλά ειδήσει. Παρ' όλα αυτά. Γιατί πάντα έρχεται και το αλλά, Υπάρχουν σοβαρέ ε, ενδείξει ότι αυτό στρεβλώνει. Τα tax rulings αυτά στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Θα ζητήσω λοιπόν ε, ενέργεια περαιτέρω ερευνών. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Κατά δεύτερον, συνεχίζονται και οι έρευνε σε ό,τι αφορά ε, τις έρευνες, ε, οι έρευνες για τις κρατικές επιδοτήσεις. Μας, ζητάει, μας ζητούν ε, οι συγκεκριτές να το εξετάσουμε το συντομότερο δυνατόν αυτό. Αλλά σα τονίζω ότι και σε ό,τι αφορά το καθεστώ των κρατικών ενισχύσεων, η ποιότητα προέχει τη ταχύτητα. Θα ολοκληρώσουμε και θα κλείσουμε τις υποθέσεις μόλις έχουμε εξαντλήσει το αντικείμενο. Τέλος, θέλουμε να δώσουμε περαιτέρω καθοδήγηση στα κράτη-μέλη και στις ε, επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις πρακτικές φορολογικού προγραμματισμού των χωρών. Για να υπάρχει σωστή καθοδήγηση θα πρέπει να επιλέξουμε καταρχάς ένα επαρκή αριθμό υποθέσεων και να αξιολογήσουμε υπό ποια μορφή θα μπορούσε να δοθεί αυτή η καθοδήγηση και πώς θα εξασφαλίσουμε την απαραίτητη σαφήνεια και για τα κρατημέλη αλλά και για τους φορείς, τους συμμετέχοντες της αγοράς. Χαίρομαι που αυτό το υποστηρίζουν οι συγητές γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη σε όλα τα επόμενα βήματα και να βελτιωθούν οι προσπάθειές μας. Του των λεχθέντων, ε, αν είπα μόνο να ακούσω τι έχετε να μου πείτε σήμερα, αλλά και τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε στο μέλλον και για τις εκθέσεις όταν θα ολοκληρωθούν, πώς θα πρέπει να αποτελέσουν και θα μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε όλες τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την Επιτροπή Φιστάκερ για την συνεκτικότατη αυτή παρουσίαση. Και τώρα να ακούσουμε τους ομιλητές. Δύο λεπτά. Σας εστίνω γιατί θα σας κλείνω το μικρόφωνο. Ο Βέρνερ Λάγκρο, ο οποίος είναι και εισηγητής για την ανταγωνισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πελφάιερ. Έχετε πλήρη αρμοδιότητα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκ επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αναμεχθεί σαν χωράφια σας. Εσείς αποφασίζετε για τα θέματα της πολιτικής αυτής. Την ελπίδα ότι θα αλλάξει κάτι στα κράτη-μέλη, την άφησα κατά μέρο σήμερα. Την ε, ελπίδα ότι θα δραστηριοποιείταν ε, διεθνώ ο Επίτροπο Μοσκοβισή, δεν την είχα ποτέ, αλλά έχω ελπίδε εναποθετημένε σε εσά. Γιατί το άρθρο 107 των Ευρωπαϊκών Συνθήκων αναφέρει ότι σε ό,τι αφορά το κινητικό δίκαιο και την, ε, το εθνικό δίκαιο, προβλέπει τα περιστρέβλωσης. Τέσσερα κράτη-μέλη λοιπόν ε, πλήττονται που έκαναν τέτοιες ε, δραστηριότητες που στραβλώνουν τον ανταγωνισμό. Στο Λουξεμβούργο έχουμε 376 τέτοιε ενέργειε που στραβλώνουν τον ανταγωνισμό. Να επαναλάβω το παράδειγμα τη Amazon. Όταν ε, χρησιμοποιώ το Amazon στην Γερμανία, πληρώνω 30% φόρο στα σύνορα εκπίπτεοφόρου και στο Λουξεμβούργο αναφέρεται ότι το Amazon ότι η Amazon πληρώνει φόρο 0,45 έως 0,55. Αυτό είναι υπέρ μια και μόνο ε, εταιρεία και αποτελεί με το παραπάνω στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εσείς είστε μοναδική ελπίδα που έχω να κινηθεί κάτι. Και όχι μόνο. Δεν τίθεται μόνο το θέμα ποιότητα, ε, τίθεται και θέμα ταχύτητα. Ένα χρόνο έχει περάσει και δεν έχω. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσά. Διακόπτει όμω ο Πρόεδρο. Κυρία Επίτροπε, έχω την εντύπωση ότι φτάσαμε όλοι πολύ αργά. Ανακαλύψαμε εξαιρετικά αργά αυτό το σκάνδαλο. Όχι μόνο η Επιτροπή για τον ανταγωνισμό και την ανταγωνιστικότητα, αλλά όλοι μας. Όλο το πολιτικό σύστημα ήρθε ενώπιον ενός κοινωνικού συναγερμού, τον οποίο σήμαναν ε, ερευνητικοί δημοσιογράφοι και ε, καταγγέλλοντες πληροφοριοδότες. Και θα πρέπει να συνταραχθούμε όλοι και να κάνουμε αυτοκριτική. Από εκεί και πέρα, πώς μπορούμε να έχουμε υγιή ανταγωνισμό όταν η φορολογική πολιτική είναι εθνική και όταν η αρχή της προσέλκυσης των επιχειρήσεων που πρέπει να είναι όλο και πιο ανταγωνιστικές επιτρέπει την ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών πολιτικών. Άκουσα τον κύριο Γιούγκερ σήμερα το πρωί και άκουσα και εσάς όταν ε, μιλήσατε και είπατε ότι κάθε χώρα έχει τη δική της ίδια φορολογική αρμοδιότητα και άρα μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες χώρες ή μπορεί ε, μεγάλες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντός της ίδιας χώρας ή μεταξύ διαφορετικών χωρών. Είμαι λοιπόν ότι η φορολογική πολιτική είναι ίδιον και επαιδείο αρμοδιότητας της εκάστοτε χώρας, ε τότε πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα και να πετύχουμε υγιή ανταγωνισμό. Δεν θα πρέπει επιτέλους να παραμερίσουμε την αρχή της φορολογικής αρμοδιότητας σε εθνικό κρατικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα. Συμφωνώ με τον κύριο Λάγκερ. Πράγματι πολλή δουλειά να γίνει. Δεν έχει φτάσει όμως η στιγμή επιτέλους μαζί με τον Επίτροπο Αρμόδιο για Οικονομικά να έχουμε μια φορολογική υπηρεσία σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ένα τμήμα, έναν οργανισμό, ένα χαρτοφυλάκιο που να ε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγες τις φορολογικές διοικήσεις και τις φορολογικές πολιτικές σε κάθε χώρα με σκοπό την όλο και μεγαλύτερη εναρμόνιση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούκες, στις εισαγωγικές σας ε, παρατηρήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Αναφέρατε κάτι εσφαλμένο. Είπατε ότι είναι καθήκον να φροντίσετε ότι όλες οι εταιρείε σε μία χώρα θα τη χάνουν ίσες και δίκαιες αντιμετώπισης. Δεν στέκει αυτό. Θα πρέπει να φροντίσετε όλες οι εταιρείε στην καθόλου αγορά να τη χάνουν ίσες αντιμετώπισης γιατί οι διεθνής ή ε, πολυεθνικές εταιρείας, ε, το εμπόριο αφορά όλη την εσωτερική αγορά συνήθως. Στις μεμονωμένες χώρες όμως της Ένωσης η πολυεθνικης εταιρειας το εμποριο αφορα ολη την είναι διαφορετική και είναι εθνική αρμοδιότητα αυτό. Πρώτη ερώτηση λοιπόν προς εσάς. Πώς θέλετε να κάνετε τη διάκριση μεταξύ του νόμιμου δικαιώματο ενό κράτου μέλου να διαμορφώνει ανεξάρτητα και αυτόνομα και χωρί συντονισμό με άλλα κράτη-μέλη το φορολογικό τη Καθεστώ και του, των ρυθμίσεων που προκύπτουν, που ε, έχουν ως αποτέλεσμα στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πώς θα ορίσετε πότε είναι κάτι παράνομο και κατά των συνθήκων αποτελεί κρατική ενίσχυση λόγω διαφορετικών προλογικών συντελεστών. Και αν δεν μπορείτε να απαντήσετε την πρώτη ερώτηση, η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξή. Τι θα κάνετε προκειμένου κάποια στιγμή να μπορέσετε να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση, προκειμένου να μπορέσουμε να ορίσουμε κάποια στιγμή τι αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση. Και στο μέλλον, τρίτη ερώτηση, θα κάνετε ένα έλεγχο, θα ξεκινήσετε έρευνα για την εξέταση των κρατικών επιδοτήσεων αν διαπιστώσετε ότι υπάρχει μεταφορά κεφαλίου της, ή μεταφορά της προλογικής ε, βάσης μιας εταιρείας σε μια άλλη χώρα, γιατί αυτό θα μπορούσε να γίνεται για φορολογικούς σκοπούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στόρβαλς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Επίτροπε Φεστάγκερ που είστε εδώ. Ένα από τα βασικά προβλήματα εδώ είναι η απουσία ενός παιχνιδιού επί ίσης όρης. Και δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε παιχνίδι επί ίσης όρης. Γιατί, γιατί οι χώρες είναι πολύ διαφορετικές, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές, χώρες περιφέρειας και χώρες στο κέντρο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επέτρεψε τη συγχώνευση δύο τηλεπικοινωνιακών εταιριών και είπατε ότι, είστε, ότι αυτές οι δύο τηλεπικοινωνιακές εταιρείες είναι δύο πολύ μεγάλοι παίκτες στη Βόρεια Ευρώπη. Είναι όμως πολύ μικροί συγκριτικά με άλλους παίκτες στην ευρωπαϊκή αγορά. Άρα τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις έδιωξε τις επιχειρήσεις, τις, αναγκα... τις ανάγκασε να περιοριστούν στην περιφέρεια. Και άρα οι επιχειρήσεις δεν είχαν άλλη εναλλακτική από το να αναζητήσουν επιθετική φορολογική πολιτική ορισμένων κρατών για να διατηρήσουν το μερίδιο της αγοράς τους. Συμπεραίνω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, δίνει κάτι με το ένα χέρι το οποίο παίρνει τελικά με το άλλο χέρι και αυτό δεν έχει καμία σχέση με το παιχνίδι επί ίσης όρης. Και όσο η Επιτροπή ε, λειτουργεί έτσι, πάντοτε θα έχουμε πρακτικές φοροαποφυγής και λαξ λίξ. Ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε στο ερώτημα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βιέγκας, ε, Πορτογάλος, καλημέρα σας. Τρεις σύντομες ερωτήσεις προς την κυρία Επίτροπο. Καταρχάς, ο κατάλογος των φορολογικών εμπειρογνωμόνων. Έχουμε των προνομιακών ε, φορολογιακών καθεστώτων. Έχουμε τέσσερα κράτη, το Λίχτενσταν μεταξύ άλλων και μικρά κρατήδια δηλαδή, ε, τέτοιου τύπου. Ε, υπάρχει πρόβλημα με την ανταλλαγή πληροφοριών. Τι μπορείτε να μας πείτε για αυτόν τον κατάλογο του ΩΣΑ, πώς μπορούν οι πολίτες να έχουν εμπιστοσύνη στις πολιτικές αν τελικά δεν κάνει τίποτα η Ευρώπη. Από εκεί και πέρα. Η έκθεση αναχώρα, το reporting, ε, ως προς την δημοσιότητα αυτών των εκθέσεων. Μιλήσατε για αξιολόγηση αντικτύπου, για μελέτη αντικτύπου. Μα ποιος θα την κάνει. Θα είναι πάλι η Price Waterhouse και Coopers Από εκεί και πέρα, η έρευνα στη Γερμανία. Είστε σε θέση να μας πείτε πόσες φορολογικές συμφωνίες θα αναλυθούν και ποιες επιχειρήσεις εμπλέκονται. Μας λέτε ότι ορισμένα ε, προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και ορισμένου τέτοιου είδου συμφωνίε είναι νόμιμε. Αφού είναι νόμιμε, τότε γιατί δεν διαδίδεται αυτή την πληροφόρηση. Δεν υπάρχει κόλλημα. Επόμενο ομιλητή. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ για τη δεσμευσή σα. Θα ήθελα να σα ε, ρωτήσω για τη μεταρρύθμιση, για την αναθεώρηση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών. Όλα τα κράτη-μέλη φαίνεται ότι πλέον συνεργάζονται με τι υπηρεσίε σα σε ό,τι αφορά τι πρακτικέ αυτέ ε, και με την έρευνα την οποία διεξαγάγεται. Μπορείτε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες για το αποτέλεσμα το οποίο θέλετε να πετύχετε, για το πώς θα αποφύγετε το φορολογικό dumping στο μέλλον. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε για να αλλάξετε τον άδικο ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών σε δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων. Θα υπάρξει εναρμόνιση οι επιχειρήσεις ε, οι οποίες ε, λαμβάνουν ε, παράνομες κρατικές ενισχύσεις θα αντιμετωπιστούν με τρόπο για να αποφευθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Πιστεύετε ότι θα πρέπει τα χρήματα αυτά να επιστραφούν στον κοινωτικό προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά τέλος τους πληροφοριοδότες. Είμαι βέβαιος ότι υποστηρίζεται μια έρευνη έρευνα για τις κρατικές ενισχύσεις. Έχει να κάνει αυτό και με την οδηγία για τους μετόχους. Το σκάνδαλο για το LuxLeaks βασίζεται και σε ό,τι αφορά πληροφοριοδότες. Ε, ο κ. Λετούρ, ε, οποίος απειλείται με φυλάκιση θα δώσετε ένα ειδικό καθεστώς για το μέλλον, για τις πληροφοριοδότες, για να τις προστατεύσουμε δηλαδή. Ευχαριστώ. James. Thank you. In considering tax competition, we... Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά το προλογικό ανταγωνισμό, να υπενθυμίσουμε ποια είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος της επιχειρήσης που θα πρέπει να είναι αγωνιστικός στο παγκόσμιο προσκήνιο, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω ένα παράδειγμα στο Ενωμένο Βασίλειο, που ήταν κορυφαίο κράτο σε ό,τι αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη στα φαρμακευτικά. Και τα τελευταία δέκα χρόνια ε, αγωνίζεται να μείνει στην πρώτη δεκάδα. Πέσει διαρκώ. Πρόκειται για μια χρόνια κατάσταση, ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο έχει να κάνει με του ευρωπαϊκού κανόνε για τι ε, ε, δοκιμέ των φαρμάκων. Γι' αυτά εκτείνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλέ εταιρείε έρευνας, όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν θέματα γιατί φοβούνται ότι θα αναγκαστούν να διεξαγάγουν την έρευνά τους εκτό τη Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να ε, ε, αντιμετωπίσουν πολύ πιο υψηλό κόστος μέσα στην Ένωση. Την προηγούμενη εβδομάδα μια άλλη επιτροπή εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια απόφαση η οποία προσθέθεσε άλλη μια πρόκληση σε αυτές που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Αυτό επηρεάζει τη συνεργασία για τις ε, προσωπικές εταιρικέ προλογίσεις. Όλα αυτά λοιπόν ξέρετε είναι αλλοσυνδεόμενα. και φυσικά και δικαιολογείται αυτά που κάνετε και έχετε αγγίξει κάποιε πτυχέ, όπω για παράδειγμα οι κρατικέ ενισχύσει και η εναρμόνιση αλλά μπορείτε κατηγορηματικά με το χέρι στην καρδιά να μα πείτε ότι θα μα δώσετε ω Επιτροπή πρόσβαση στα έγγραφα αυτά και στι προτάσει τι οποίε εξετάζετε γιατί το παράδειγμα του σημερινού πρωινού είναι ότι η Επιτροπή λαμβάνει μία απόφαση χωρίς να έχει ουσιαστικά όμως επαφή και με τους υπόλοιπους φορείς. Γίνεται λίγο ξεχωριστά Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάπελ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επιτροπέ. Από το σχέδιο της έκθεσης Φεραϊρά και τώρα φαίνεται ότι η υπηρεσία σας από το 99 έχει ερευνήσει 95 ε, υποθέσεις φορολογικής ε, αποφυγής και τώρα τέσσερις υποθέσεις εξετάζει σε ό,τι αφορά και το LuxLeaks. Και εδώ πέρα αναφέρεται και η πτυχή των κρατικών ενισχύσεων. Το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της έκθεσης ε, Φέρμπερ επιθυμούν αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από το 2016 και μετά, από το 2016 και μετά. Όχι μόνο ανταλλαγή διασυνοριακών πληροφοριακών, αλλά όλων των φορολογικών αποφάσεων. Και αυτό μάλιστα με αναδρομική ισχύ 10 ετών. Μπορείτε να μας ε, μπορείτε να μας πείτε αν υπολογίζετε ότι θα προκύψουν πολύ πιο πολλές υποθέσεις έρευνας με τη μεγάλη εισρωή αυτών των δεδομένων. Έχετε τους πόρους αυτούς να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά και κάτι άλλο στο θέμα έκθεσης ε, Φεραίρα και Τόιρερ. Προτείνεται να υπάρξει μεσοπρόθεσμα ένα σημείο εγκαθάρισης και ενδεχομένως αυτό να βρίσκεται στα πλαίσια της υπηρεσίας σας. Πώς τοποθετήσετε ένα άλλο θέμα από το σχέδιο έκθεσης. Δεν προκύπτουν όλα τα κράτη-μέλη. Μάλλον ότι δεν ανταποκρίθηκαν όλα τα κράτη-μέλη στην υποχρέωση χορήγηση δεδομένων και η δική μου η χώρα, η Αυστρία. Αυτά βέβαια μέχρι 20 Ιουλίου. Μέχρι 20 Ιουλίου μα είπατε ότι εδώ μεταξύ, στο μεταξύ διάστημα συνεργάζονται όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Έστω Yes, thank you. I'd like to talk to you. Ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη σχέση ανάμεσα στις αναχώρα εκθέσεις και τη δική σας εργασία, εργασία σας εσά και των υπηρεσιών σας. Πώς η αναχώρα έκθεση θα σας βοηθήσει στο να καθορίσετε τη νόμιμη χρήση των κρατικών επιδοτήσεων ή ενισχύσεων, τι είδου σύστημα πρέπει να συμπληρώσουν ώστε εσείς να μπορείτε να λειτουργήσετε, δημόσια ή μη δημόσια ε, κριτήρια και έπειτα από την άλλη πλευρά πώς ε, ε, θα έπρεπε να φτιαχτεί αυτό το σύστημα ώστε να μην είναι σε μειονεκτική θέση ευρωπαϊκές εταιρείες σε, όταν αυτές συναγωνίζονται με εταιρείες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τζάνι. Ευχαριστώ πολύ. Κάποτε καταλαβαίνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφορες ε, επιτροπές και τα κεντρικά ζητήματα είναι τα τυπικά ή που θα μπορούσαμε να τα πούμε τυπικά. Ε, απάντως υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να βρεθούν μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Για να είμαι πολύ συγκεκριμένος και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα που μπορεί να είναι επίσης χαρακτηριστικό. Ας πούμε στη χώρα μου, την Ουγγαρία, η Ουγγρική κυβέρνηση δημιουργεί, δημιουργεί συγγνώμη, κατασκευάζει ένα νέο πυρηνικό εργοστάσιο φυσικά με τα χρήματα των φορολογούμενων. Σύμφωνα με τις ε, τρέχουσες εκτιμήσεις, ε, η τιμή του ηλεκτρισμού θα φτάσει στα ύψη. Αυτό θα καθορίσει όμως και όλο την υπόλοιπη όλες τις τιμές των διαφόρων ε, προϊόντων. Δηλαδή τελικά τα χρήματα των φορολογόμενων επενδύονται σε ένα σύστημα το οποίο θα υψώσει τις τιμές γενικά, τις τιμές της ενέργειας καταρχήν και στη συνέχεια των υπολείπων. Και όλο αυτό γίνεται μέσω, σε παρενθέσεις, μέσω ε, ε, ε νόμιμων μέσων, αλλά είναι σίγουρα κατά κάθε ε, Αρχή της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης. Πώς μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να λύσουμε τέτοια προβλήματα και τέτοιες καταστάσεις. Ευχαριστώ. Έχω και μια ερώτηση από το Κατσιδιάη. Μόνο για έναν έχουμε χρόνο. Η κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν βρίσκεται ε, χρήσιμες τις αναχώρα εκθέσεις και κατά πόσο θα έχουμε υποχρέωση ε, με βάση την οδηγία περί ε, ε, λογιστικών ελέγχων για το κατά πόσο έχει δοθεί κάποια προτιμησιακή, κάποιο προτιμησιακό φορολογικό καθεστώς στην λόγω εταιρείε και αν υπάρχει και προστιθέμενη αξία για αυτές. Σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε. Σας ευχαριστώ πολύ. για την ερώτησή σας. Για τις ερωτήσεις σας. Καταρχήν. Καταρχάς να αρχίσω από την αρχή. Λοιπόν, Βέρμαν, δεν έχω χάσει τις ελπίδες μου, όχι. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μου, αλλά και σε εσά. Αλλά και στα κράτη-μέλη. Ότι θα πράξουν το σωστό. και νομίζω πως θα πρέπει να κατευθυνθούμε από το αίσθημα των ε, πολιτών ότι δεν είναι δίκαιη αυτή η κατάσταση. Κάναμε διάφορα πράγματα και προσπαθούν στη διάρκεια της κρίσης να εκτίσουν τον έλεγχο των προπολογισμών τους. Είδανε τις τιμές να ε, πέφτουν, α, τους μισθούς να πέφτουν και να μένουν ότι οι εταιρείε δεν θα, χάσουν ούτε πολλά ούτε λίγα, αλλά το, αυτό που τους αντιστοιχεί και αυτό είναι το δίκαιο. Άρα οι πολίτες περιμένουν από εμά να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ούτε μια εταιρεία δεν θα κερδίσει ή δεν θα έχει προτιμησιακή μεταχείριση ε, η οποία δεν θα προσφέρεται και στις υπόλοιπες εταιρείε. Νομίζω ότι είναι βάσιμη αυτή η ελπίδα γιατί πιστεύω πως είναι κοινή αυτή η στόχη για όλους μας και σε αυτό βεβαίω δουλεύουμε όσο γίνεται ταχύτερα. Για το θέμα του πώς μπορούμε να μιλήσουμε για ισότιμο όρος του παιχνιδιού όταν υπάρχουν τόσες διαφορές. Καταρχήν πιστεύω ναι, πως για μένα ή ε, θεωρώ ότι η συνθήκη είναι κάτι το δεδομένο. Διότι έχουμε έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, έχουμε τη δυνατότητα επιβολής της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Δεν είναι η ζούγκλα, δεν είναι λεσεφέρ, δεν είναι ο, αυτός ο στόχος μας. Η συνθήκη λέει ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτού του περιορισμού. Αλλά ακόμα και αν έχουμε τα ίδια φορολογικά ποσοστά, πάλι θα υπάρχουν διαφορέ όταν κάποια εταιρεία ε, θα αποφασίζει πού θα τοποθετήσει την έδρα τη, πού θα τοποθετήσει το ερευνητικό τη τμήμα και ούτω καθεξής. Γιατί υπάρχουν πάντα διαφορέ στι υποδομέ, ε, στα δεξιότητε, στα προσόντα των ε, πιθανών εργαζόμενων, πόσο στενά θα συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια κτλ. κτλ. Δεν θα πρέπει να προσπαθούμε λοιπόν να πετύχουμε το αδύνατον και να τα εξομοιώσουμε όλα. Γιατί εξακολουθεί να είναι υγιές το να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά όχι ο αθέμητος. Ακόμα όμως και για την επίτευξη αυτού έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά. Το αίτημα για έναν καθαριστικό ε, οίκο, ε, για μια νέα αρχή. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε. Γιατί ε, πιστεύω πως ο κώδικας διοντολογίας και ο ΩΣΑ κάνουν καλή δουλειά. Στο σχέδιο PEPS για τη διάβρωση βάσης και, μεταφοράς, και τη μεταφορά κερδών κάνουν σωστή δουλειά για να ελέγξουν σε μεγαλύτερο κλίμακα από ότι της Ένωσης γίνεται στο πλαίσιο του ΟΣΑ γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί έχει, έχει οδηγήσει σε πρόοδους. Για να σας δώσω και κρυμμένο παράδειγμα της πρόοδου που έχει σημειωθεί, όταν, όταν μιλάμε για τα, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ας πούμε, και τα σχετικά τις σχετικές διατάξεις. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τόσα αν είχαμε ακολουθήσει μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε μια αναπογραφή των όσων έχουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε πριν αρχίσουμε να προσπαθούμε να φεύγουμε κάτι νέο. Γιατί κάτι τέτοιο θα μας πάρει πολύ χρόνο να το καταφέρουμε. Και το θέμα των σχετικών αγορών. Πιστεύω όταν ε, τουλάχιστον ε, ασχολήθηκα με το τομέα του ανταγωνισμού, ήταν εντυπωσιακό που είδαμε ότι μπορεί να υπάρχουν παγκόσμιε εταιρείε, αλλά πολύ εθνικέ αγορέ. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε ας πούμε για το ότι έχουμε ας πούμε τα τηλέφωνα τα τηλέφωνα, ενώ είναι τεράστιες εταιρείε παγκόσμιου κλίμακα, έχουμε πολύ συγκεκριμένες εθνικές αγορές. Και γι' αυτό και μιλάμε για ψηφιακή αγορά, έτσι ώστε να είναι ευρύτερη, μεγαλύτερη αγορά, ώστε οι εταιρείε να μπορούν να αναπτυχθούν καλύτερα και να ανταγωνίζονται άμεσα μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα παράδοξο βέβαια, γιατί μιλάμε για την ενιαία αγορά εδώ και δεκαετίες και σε ορισμένου τομεί λειτουργεί εδώ και δεκαετίες και έχει εξυπηρετήσει τα πράγματα. Όμως στον ψηφιακό τομέα δεν έχουμε ενιαία ψηφιακή αγορά. Δεν έχουμε μια ενεργειακή αγορά, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να την αποκτήσουμε, να τις αποκτήσουμε. Εργαζόμαστε πολύ εστιασμένα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα αλλάξουμε ή δεν θα μετακινήσουμε το σύνορο για το τι είναι φορολογία και τι είναι νομοθεσία, για τα κράτη-μέλη και τι είναι έλεγχος των κρατικών ανισχύσεων. Και άρα εκεί έχουμε πολύ σαφή κριτήρια, ώστε να μπορούμε να έχουμε αυτή τη διάκριση για το πότε και πού παρεμβαίνουμε στις εθνικές αρμοδιότητες και πότε κάνουμε αυτό που μας επιβάλλει η συνθήκη, ότι δηλαδή να εξασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχει παράνομη ή ασύμβατη φορολογική βοήθεια. Και, εδώ, και γι' αυτό έχουμε κριτήρια εμπορικά, επιλεξιμότητας και ένα σωρό άλλα κριτήρια, γιατί διαφορετικά θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Ορισμένα από αυτά τα κριτήρια βεβαίως μας επιτρέπουν επίσης να έχουμε μια ενημερωμένη αξιολόγηση όσον αφορά τη μεταφορά των κερδών με χρηματοπιστωτικά ε, μέσα, συμφωνίες τιμών και άλλους τρόπους μεταφορών, μεταφοράς κερδών. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν μηχανισμό που δεν παρεμβαίνει στις εθνικές ε, ε, αρμοδιότητες για να αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσει η φορολόγηση των εταιριών και των ομίλων. Αυτό εν μέρει νομίζω απαντά και στο κύριο Τόρβαλς ε, για το ισότιμο πεδίο κανόνων το έχουμε, ακόμα και αν έχουμε μεγάλες εταιρείες που θα είναι ενεργές σε 4, 5, 10, 15 κράτη-μέλη. Έχουμε ωστόσο ε, εθνικές αγορές και γνωρίζετε ότι στην εντολή μου έχω τρία διαφορετικά να κάνω. Έλεγχο κρατικών ισχύσεων, έλεγχο συγχωνεύσεων και αντιτράστ. Και έλεγχος μονοπωλίων. Όταν ελέγχουμε τι συγχωνεύσει, εμεί δεν αναμειγνιόμαστε στι ε, ε, εταιρικέ αποφάσει. Απλώ πρέπει να ελέγξουμε αν μια τέτοια απόφαση θα στρεβλώσει ή θα φημώσει τον ανταγωνισμό, γιατί ο ανταγωνισμός προσφέρει στους καταναλωτές ε, μεγάλο φάσμα τιμών, καλή ποιότητα και καινοτομία. Αλλά δεν νομίζω ότι για οποιαδήποτε εταιρεία, ό,τι και αν γίνει στον έλεγχο συγγονεύσεων, μπορεί κάτι τέτοιο να αποτελέσει δικαιολογία ώστε να αναζητήσει ε, κέρδη μέσα στο το φορολογικό σύστημα. Αυτό είναι τελείως διαφορετική υπόθεση. Για το θέμα του κύριου Μαραγκέλ, είναι, για το θέμα των τρίτων χωρών, είναι κάτι διαφορετικό, γιατί βέβαια οι τρίτε χώρε είναι εκτό του δικού μα ελέγχου. Όταν όμω πρόκειται για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για το προσωπικό εισόδημα, εδώ έχουμε αποτελέσματα. Γιατί οι διαπραγματεύσει με τρίτε χώρε μα επέτρεψαν κάποια πρόοδο, ώστε να μπορέσουν και εκείνοι να ανταλλάσσουν πληροφορίε μαζί μα. Ανοιχτή λοιπόν και διάφανη ε, διαγωνισμοί, προσφορές όπως έγινε με την Price House Coopers. Γι' αυτό και ζητάμε από το κάθε κερδός να μας δώσει 10 με 12 συγκεκριμένες φορολογικές εξαιρέσεις ή προνομιακές φορολογήσεις για να δούμε πώς αυτά τα tax rulings τα επωνομαζόμενα, λειτουργούν στα λόγο κράτος. Δεν δημοσιεύουμε τα ονόματα των λόγω εταιριών διότι από την αρχή μέχρι, τις, ε, μέχρι το τέλος αυτής της ανάλυσης δεν έχουμε εκ των προτέρων λόγο να, να, να, πιστεύουμε ότι έχουν κάνει κάτι στραβό και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη ώστε να μεριμνήσουμε καμιά εταιρεία να μην κατηγορείται αδίκως για ατυπίες ή αντικανονικές συμπεριφορές. Δεν έχω ε, δε, κάποια συγκεκριμένη ιδέα για το πώς θα διευκολύνεται η αναχώρα έκθεση αναφορά. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να έχουμε ε, διάφανη ματιά στη πραγματικά φορολογικά ποσοστά γιατί αν μηδενιστούν σε μια χώρα τότε βεβαίω είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι απόδειξη ενός ωφέλους που οφείλεται σε φορολογική βοήθεια. Αυτό θα διευκόλυνε τη δουλειά μας. Δεν ξέρω τώρα αν και πώς λειτουργεί ο φαρμακευτικός τομέας και γι' αυτό και δεν μπορώ να σας σχολιάσω. Να σας το σχολιάσω. Πάντως, ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία για τη συζήτηση για το μέλλον είναι τα κοιτία ε, αυτά των ε, ε, ευρεσιτεχνιών, γιατί αυτό αποδεικνύει πως γίνεται έρευνα και ανάπτυξη στο κάθε κράτος μέλος και να αναγνωρίζεται κατά αυτόν τον τρόπο η επένδυσή σου. Αντίθετο με το, το, το, λογικό καθεστώς που είναι ευνοϊκό για τις ευρεσιτεχνίες και το εκμεταλλεύεται κανείς μόνο και μόνο για να έχει όφελος φορολογικό. Όχι για να επενδύσει ε, στην ευρεσιτεχνία την ίδια. Είναι καλό να προωθηθεί δηλαδή η έρευνα και η ανάπτυξη και η ευρεσιτεχνία αλλά όχι η χρήση αυτής μόνο και μόνο για φορολογικούς σκοπούς. Τώρα, η DG ότι εγώ δεν θα πρέπει να έχουμε και τους πόρους να ελέγξουμε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό το οποίο θα έπρεπε να έχουμε είναι η δυνατότητα να ε, ελέγξουμε όταν έχουμε υποψίες ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί τα κράτη-μέλη πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και να έχουν συστήματα φορολόγησης που να ε, λειτουργούν σε πλήρη συμφωνία με τον κανονισμό τους περί κρατικών ενισχύσεων. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορούμε να πάμε στη ρίδα του θέματος, όχι ακόμα έχουμε όλα, γιατί αλλιώς δεν προλαβαίνουμε παρά μόνο ελέγχουμε. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε και στην πηγή του προβλήματος και να μπορέσουμε να δώσουμε και κατευθύνσεις. Και κάνω μια διάκριση όταν αφορά ε, συγκεκριμένες δράσεις ή κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να μας πάρει περισσότερο καιρό το να καταλήξουμε σε κατευθυντήριες γραμμές που έχουν και πιο δεσμευτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρούμε τρόπο να δώσουμε κατευθύνσεις μέσα σε πιο προβλέψιμο χρονικό πλαίσιο για να μπορούν τα κράτη-μέλη να δουν ποια είναι η καλύτερη πρακτική, πώς μπορούν να γίνουν τα πράγματα, πώς μπορεί να προλάβει τα προβλήματα τέτοιου τύπου που τα δείχνουν και οι εκκρεμείς υποθέσεις που εξακολουθούμε να έχουμε. Για το θέμα το, της Ουγγαρίας, επίσης είναι έρευνα για κρατικές ενισχύσεις, όχι για φορολογικά θέματα ή δημοσιονομικά θέματα. Ε, ε εδώ Έχουμε διάφορες ερωτήσεις να θέσουμε στις Ουγγρικές Αρχές για το ακριβώς πώς χρηματοδοτείται αυτό το έργο, για αν υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις, ε, όπως αυτό που, αυτές που είπατε στην ερώτησή σας. Η δημόσια διαβούλευση για τις αναχώρες εκθέσεις ελπίζω να μας φέρει σε ένα σημείο που θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σύντομα, γιατί από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμή είναι ακριβώς η μετακίνηση κερδών από τη μια χώρα στην άλλη και η παρακολούθηση αυτού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια για τις αναχώρα εκθέσεις. Ελπίζω λοιπόν ότι θα φτάσουμε σε κάτι τέτοιο και θα βρούμε έναν τρόπο ώστε να είναι όλα αυτά ισορροπημένα. Πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Παράδειγμα είναι και πώς γίνονται τα πράγματα στην ΣΥΠΑ, γιατί σε ορισμένους τέτοιους τομείς έχουν περισσότερη ε, διαφάνεια. Και από ό,τι φέρονται, οι επιχειρήσεις τους ε, ευημερούν. Ίσως θα πρέπει από αυτούς να εμπνευστούμε λοιπόν για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα πράγματα, για να έχουμε σωστή ισορροπία. Γιατί βεβαίως ποτέ δεν θα πρέπει να φτιάχνουμε έναν κανονισμό ο οποίο να είναι βάρος για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να εξισορροπεί τα αποτελέσματα, ότι δηλαδή κάθε εταιρεία που το κάνει, λειτουργεί σωστά, θα ξέρει ότι ε, θα μπορεί να έχει κάποια φοροαπαλλαγή, ας πούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την Επίτροπο Φεστάγκερ. Πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Να δώσω την Προεδρία τώρα στον Αλάν Λαμασούχ για τις καταληκτικές του παρατηρήσεις και για πρακτικές ανακοινώσεις. Παρακαλώ, Αλάν. Ευχαριστώ πολύ, Ρομπέρτο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο γιατί απάντηση συγκεκριμένα σε όλες τις ερωτήσεις όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι δείξατε ότι Πέρα από τις υποθέσεις οι οποίες ε, είναι υποδιερεύνηση αυτή τη στιγμή και για τις οποίες μας είπατε ότι τελικά θα γίνουν πολύ πιο πολλοί άριθμες από ό,τι θα φανταζόταν κανείς, μέσα από τις διαδικασίες και τους κοινοτικούς κανόνες κατά των κρατικών ενισχύσεων συμβάλλατε στη δημιουργία πολιτικής πίεσης και άσκηση ε, αυτής έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να δεχθούν να μπει ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές και να καταφέρουν σε βάθος χρόνου, σε εύθετο χρονικό ε, διάστημα, να εναρμονίσουν τον ορισμό των φορολογητέων κερδών. Και αυτό είναι στόχος δικός μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τούτων λεχθέντων. Ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως και εμείς και εσείς είναι το follow-up, η παρακολούθηση. Να προσπαθήσουμε να είμαστε σε εγρήγορση, να παρακολουθούμε την κατάργηση μη φυσιολογικών πρακτικών, να παρακολουθούμε την τροποποίηση σκανδαλωδών πρακτικών, να ε, παρακολουθούμε όταν γίνεται αυτό βάσει των εντολών του ΩΣΑ να μην ξαναμπαίνει, όταν φεύγει από την πόρτα, να μην ξαναμπαίνει από το παράθυρο με κάποιο άλλο τρόπο. Είδαμε το pattern box, το κοιτίο διπλωμάτων έβρεση τεχνίας, το οποίο τελικά αντικαταστάθηκε από το <clears throat> κουτί από το κοιτίο καινοτομία. Ό,τι έχει θετικό αποτέλεσμα και τροποποιεί την εθνική νομοθεσία είναι καλό. Έχουμε δει όμως ότι ψηφίζονται αυτά, εφαρμόζονται αυτά και τελικά ξαναπροκύπτουν τα θέματα με, ενδεδημένα με άλλη μορφή μετά από 5-10 χρόνια. Ευχαριστώ όλους. Ο Πρόεδρος ευχαριστεί ευγενικά και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Σας ευχαριστώ που διοργανώσατε και ήσασταν παρόντες σε αυτή ε, την συνεδρίαση η οποία ήταν εξαιρετικά σημαντική και νομίζω ότι δεν μας απογοήτευσε. Ευχαριστώ.